Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας πρωινή συνεδρία. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς τα εξής. Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Βελγίου, ο κύριος Ντάνι Πίτερς, έχει ανελημμένες υποχρεώσεις διότι διεξάγονται, όπως γνωρίζετε, ε, διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετούς μήνες στη χώρα του Βελγίου για το θέμα της κυβέρνησης. Και ο κύριος Μάγερς, αντιπρόεδρος της Γερουσίας, θα είναι εδώ μαζί μας και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά γιατί προσφέρθηκε θελαντικά να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Πίτερς. Θα είναι συμπρόεδρος λοιπόν με τον υποφαινόμενο στην πρωινή μας συνεδρία, η οποία θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. όχι μόνο λόγω του περιεχομένου αυτών που θα συζητήσουμε, αλλά και κυρίως χάρη στις πολύ λαμπρές προσωπικότητες που θα είναι μαζί μας και θα συμμετέχουν στο σχολιασμό και θα μοιραστούν μαζί μας τους προβληματισμούς τους. Καταρχάς λοιπόν, να ακούσουμε τις ε, παρουσιάσεις των εκθέσεων των ομάδων εργασίας. Οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν χθες. Και εάν δεν έχετε λάβει, θα λάβετε εντός ολίγου το έντυπο το οποίο θα συμπληρώσετε για να ζητήσετε το λόγο στη συνέχεια μετά την παρέμβαση του Προέδρου του, Προέδρου του Συμβουλίου, του κύριου Ιβ Πρωθυπουργού του Βελγίου και μετά τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Μπαρόζο. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι πρόθεσή μου είναι η εξής. Όταν καταρτιστεί ο κατάλογος των παρεμβενόντων, να φανεί ποιοι είναι οι συνάδελφοι που επιθυμούν πραγματικά να λάβουν το λόγο για να μην έχουμε ένα πολύ μακροσκελή κατάλογο. Δηλαδή από την αρχή της συζήτησης να ξέρουμε πόσοι θέλουν το λόγο. Θέλουν 10 ή θέλουν 50 το λόγο. Καλώς για να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα το χρόνο και να δώσουμε ε, το χρονικό περιθώριο στον καθένα να πάρει το λόγο και να εκφραστεί. Αυτά για αυτά τα θέματα τα διαδικαστικά. Να περάσουμε στις παρουσιάσεις των εκθέσεων των εισηγητών ε, στις ομάδες εργασίας. Να δώσω το λόγο καταρχάς στον εισηγητή της ομάδας εργασίας υπαριθμών 1, μια ομάδα εργασίας η οποία ασχολήθηκε με το είδος ανάπτυξης και το είδος θέσεων απασχόλησης που επιθυμούμε για την Ευρώπη αύριο. Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ήταν ο συνάδελφος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 Κάναμε μια σύντομη εισαγωγή. Σε αυτή την εισαγωγή εγώ είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στα μέλη της ομάδας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της στρατηγικής για το 2020 και βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2011 και γι' αυτό στη συνέχεια όλοι πήραν το λόγο και συμφώνησαν στο ότι η ανάπτυξη θα λάβει χώρα μόνο μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής, μεγαλύτερης παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική ατζέντα. Επίσης υπέβαλα και κάποιες ιδέες στην ομάδα εργασίας για να αναζωπυρώσω τη συζήτηση ακόμα περισσότερο. Μιλούμε λοιπόν για την πράσινη οικονομία, για την, για την οικονομία της γνώσης και για την πράσινη έρευνα. Μιλούμε επίσης για τη συμμετοχή των νέων, αλλά και για τον, τη συμμετοχή των μεγαλύτερων, μεγαλύτερης ηλικίας στην παραγωγική διαδικασία. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τονίσουμε. Θα πρέπει να εγγυηθούμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία οφείλει να διαδραματίζει ρόλο κλειδί στις εξελίξεις. Όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας πήραν το λόγο και τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μείωση ε, δημόσιου χρέους από τη μία, χωρίς όμως να αποτελέσει αυτό τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη από την άλλη. Βεβαίως πρέπει η Ευρώπη να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση, να ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη, μειώνοντας τα ελλείμματά της. Η μείωση του δημόσιου ελλείμματος ουσιαστικά ε, σημαίνει και, και λαμβάνει χώρα μόνο μέσω της καλύτερης διαχείρισης των δαπανών. Ε, και ελοχεύει ο κίνδυνος η κρίση να μονιμοποιηθεί. Και αυτό θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Ζητούμε λοιπόν όντως τη μείωση των δημοσίων ελλημάτων, όμως πρέπει να έχουμε καλύτερη κατανομή των οικονομικών δυνάμεων και των εργαλείων προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει δηλαδή ε, το μισθολογικό βάρος να ελαφρυνθεί για τους ε, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ε, τονίσαμε επίσης ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν μόνο ως στόχο πολύ συχνά το βραχυπρόθεσμο κέρδος και πολύ συχνά είναι παρούσες για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη χώρα. Από την άλλη, ε, ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνάει ολόκληρο και ΑΕΠ ολόκληρης χώρας πολύ συχνά. Γι' αυτό και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να τις καλέσουμε και να τους επιβάλλουμε να αναλάβουν πολύ περισσότερη και πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη. Να αλλάξουν οι νοοτροπίες στις ηγετικές θέσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να διευκολύνουμε και την πίστοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη. Και θα πρέπει να στηρίξουμε την απασχόληση των νέων όσων είναι άνω των 50 ετών αλλά και των μεταναστών. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά θεωρούμε ε, ότι καταρχάς βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει περάσει η κρίση. Τα κράτη έχουν κύριο μέλημα τη σταθερότητα και λιγότερο μέλημα έχουν την ανάπτυξη. Και έτσι επενδύουν λιγότερο στην έρευνα, λιγότερο στην ανάπτυξη και η Ευρώπη χάνει σε ανταγωνιστικότητα. Και αυτό βεβαίω είναι από απειλή για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτή είναι μια διαπίστωση γενικότερα. Η εσωτερική αγορά έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από το 1992 και μετά. Αυτό έχει συμβάλει στη δημιουργία τριών εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης. Το 2008 η χρηματοπιστωτική κρίση ουσιαστικά τάραξε, συντάραξε τα θεμέλια αυτής της αισιόδοξη προοπτικής και τα βασικά βήματα της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν έλαβαν χώρα τελικά. Οι αρχές δεν έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Δεν μπορεί το κράτος από μόνο του να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ικανές και αρκετές λόγω του δημοσίου χρέους. Θα πρέπει λοιπόν οι θέσεις απασχόλησης να προκύψουν από άλλους τομείς και γι' αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν ένα συγκεκριμένο περιθώριο ελιγμών, να έχουν δυνατότητες. Αυξημένα ποσοστά ανεργίας άλλωστε σημαίνουν και μειωμένη κατανάλωση. Γι' αυτό και πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά απασχόλησης κυρίως στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που είναι δηλαδή οι νέοι και όσοι είναι άνω των 50 ετών. Αυτές οι ηλικιακέ ομάδες, οι πληθυσμιακές ομάδες έχουν πολλές δυνατότητες και μπορούν να χρησιμεύσουν στις επιχειρήσεις. Άλλωστε, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να στοχεύει καταρχάς στους Ευρωπαίους πολίτες και στη συνέχεια ε, θα μπορεί να καλεί ε, πολίτες τρίτων χωρών. Η καινοτομία είναι η λέξη κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η καινοτομία είναι αυτή που θα οδηγήσει στη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Τα μέλη της ομάδας εργασίας υπογράμμισαν ότι η αυτοματοποίηση και η ρομποτοποίηση ουσιαστικά πλήττει τις πιο, ε, τα πιο ευπαθή, αν θέλετε, επαγγέλματα, τις εργασίες που χρειάζονται τις λιγότερες δυνατές ε, δεξιότητες. Θα πρέπει να φροντίσουμε τον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Εκεί χρειάζονται συγκεκριμένες ειδικότητε και θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό, καθώς και στον τομέα της πράσινης ε, ενέργειας. Να δημιουργήσουμε λοιπόν θέσεις απασχόλησης στην οικονομία της γνώσης και στην πράσινη οικονομία. Από εκεί και πέρα τα μεγάλα έργα υποδομής μπορούν να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά και να αναζωπυρώσουν και την ανάπτυξη αλλά και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Καλύτερη κατάρτιση θα οδηγήσει σε καλύτερη απασχόληση και γι' αυτό πολλοί συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας μας έχουν εφιστήσει την προσοχή στην αναγκαιότητα της διαβίου μάθησης. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να καταρτίζει καλύτερα τους εργαζόμενούς της και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ενθαρρύνονται ώστε να παραμείνουν στην Ευρώπη, να παραμένουν και να προσφέρουν εδώ. Οι πολιτικές που θα οδηγούν στην πράσινη οικονομία θα πρέπει να είναι καλά συντονισμένες μεταξύ τους και να μην οδηγήσουν τελικά σε διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η πράσινη οικονομία θα λειτουργήσει ε, θετικά προς την συνοχή και δεν θα πρέπει να ε, συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Ένα μέλος της ομάδας εργασίας επίσης ε, παρατήρησε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ε, δεσμεύσεις όχι μόνο από πλευράς πολιτικών αλλά και από πλευράς επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα και η ομάδα εργασίας μας δούλεψε πολύ αποτελεσματικά. παρόλο που πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν παρόντα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων σε άλλες ε, επιτροπές. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις επιχειρήσεις και να δούμε τι είδους νέες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν και τι είδους καινούργιες θέσεις απασχόλησης. Τώρα, ως προς το δεσμευτικό χαρακτήρα της στρατηγικής του 2020 της Ευρώπης για την ε, απασχόληση και για την οικονομία, οι εξή ιδέες έχουν προταθεί. Τα μέλη της ομάδας εργασίας τόνισαν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ενημερώσουν τους πολίτες για τα μεταρρυθμιστικά σχέδια βάσει της καινούργιας στρατηγικής για το 2020. Άλλα μέλη της ομάδας εργασίας δήλωσαν ότι προβλήματα ανάπτυξης και απασχόλησης θα πρέπει να επιλύονται ε, με τρόπο συνολικό ε, και συλλογικό και γι' αυτό χρειάζονται κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες. Συνεργασία στο θέμα της έρευνας, της ανάπτυξης, της βιομηχανίας, ε, της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Βασικά αγαθά, βασικά προϊόντα από τρίτες χώρες μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τις προσταγές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ούτε τους κανόνες τους περιβαλλοντικούς και τους οικολογικούς. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαλέσει τα κράτη αυτά σε διεθνή φόρουμ ε, προκειμένου τα προϊόντα τους να πληρούν τις σωστές προϋποθέσεις. Έχουμε την, το επιχειρηματικό πνεύμα, την ευελιξία, την κοινωνική διάσταση, την ποιότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι ένα απόσπαστο μέρος των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί ως πρότυπο για τις ε, υπόλοιπες και τρίτες χώρες. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της πρώτης ομάδας εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Καταρχάς, σεβαστήκατε και το χρονικό περιθώριο που είχατε στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ για αυτό. 5 με 10 λεπτά έχει ο κάθε εισηγητής. Περνάμε τώρα στον εισηγητή της δεύτερης ομάδας εργασίας. Η δεύτερη ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με το είδος της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης που επιθυμούμε για την Ευρώπη αύριο. Η συνάδελφός μας, η κυρία Περβάνς θα είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας αναφέρω τις εργασίες της ομάδας εργασίας 2 για την οικονομική διαχείριση, διακυβέρνηση. Αυτή η ομάδα εργασίας ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλησα να ακολουθήσουμε κάποιες προτάσεις ισχυρές που κάναμε στην αρμόδια επιτροπή για, το θέμα της οικονομικής κρίσης. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μια σύνθεση για τα θέματα που αφορούν την Ευρώπη τη ζώνη του ευρώ, οπότε θεσπίσαμε την ομάδα Αντιπροέδρου για αυτά τα θέματα και η ομάδα μας ήδη ξεκίνησε να συζητάει το θέμα του πολέμου των νομισμάτων και αποτελεί νομίζω μια πρόοδο σημαντική ενοιολογικά. Η δεύτερη ισχυρή πρόταση που έχουμε είναι η διάθρωση μεταξύ πολυμερού επαγρύπνηση και του συμφόρου Σταθερότητα. Για να μην δηλαδή ποια είναι η καλή, η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο σημείων όσον αφορά τι τωρινέ συζητήσει. Και ένα τρίτο θέμα που αναφέρθηκε είναι ε, η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που η Κομισιόν ή το Συμβούλιο θα θέλει να εφαρμόσει στα πλαίσια της των συζητήσεων που κάνουμε. Θα ακούσετε από αυτά που είπα συναδελφοί ότι έχουμε και θέματα φορολογίας τα οποία γίνονται όλο και πιο σημαντικά στις συζητήσεις που κάνουμε οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε εδώ αναρμονικά για όλα αυτά τα θέματα. Στι άλλε παρεμβάσει και μιλίε των συναδέλφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια και των συναδέλφων των Ευρωβουλευτών θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε πέντε σημεία. Πρώτο σημείο που ήταν αρκετά επίμαχο ήταν το Ευρωπαϊκό Εξαμήνο και ο συσχετισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών εργασιών και των υπολείπων. Βεβαίως ανέφεραν οι ευρωβουλευτές τις συνθήκες υπό τις οποίες το σύνολο των προτάσεων του πακέτου που υπάρχει σήμερα θα υιοθετηθούν και πολλοί βουλευτές από την Ιταλία, τη Τσεχία, τη Γαλλία και αλλού αναφέρθηκαν στις προθεσμίες που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια για να συμμετάχουν στη διαδικασία αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η συμβολή του Εθνικών Κοινοβουλίων θα μπορούσε να περιληφθεί, να ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό το είπε ιδιαίτερα και ο Γάλλος εκπρόσωπος, ζητώντας ότι μετά την υιοθέτηση εθνικών προγραμμάτων σύγκλησης θα πρέπει να βρεθεί μια μορφή συνέλευσης ή κάποιες άλλες κοινοβουλευτικής συνεδρίασης που θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια Ενό διαγράμματος που θα γίνει περίπου το Μάιο, αλλά τέλο πάντων θα συζητηθεί περαιτέρω. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του εθνικού χρέους και ε, των ε, εθνικών ομολόγων. Το ανέφεραν αυτό οι Βρετανοί συνάδελφοι. Και ο Ιταλός συνάδελφός μας ε, αναφέρθηκε επίσης στους δείκτες όσον αφορά την βιωσιμότητα των, ε, διεθνών, το, των ε, δημοσίων οικονομικών. Ένα άλλο θέμα που συστήθηκε επίσης κατά πολύ σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα είναι το θέμα της ενδεχόμενης αναθεώρησης των συνθήκων. Οι συνάδελφοι του Προκοινοβουλίου καταρχήν ανέφεραν τις προτάσεις του Ζαγκλόρ Γιούγκερ που λέει ότι αυτή η αναθεώρηση θα ήταν απαραίτητη παρά μόνο για πολιτικούς λόγους που σχετίζονται μόνο με το, τις αποφάσεις του ΤΑΔΙ Δίνα Εθνικού Δικαστηρίου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο ενδεχομένω, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο ποτέ, θα έπρεπε να γίνει μια προστευμένη διαδικασία ή θα έπρεπε αντίθετα να διοργανωθεί μια συνέλευση και αυτό αφαιρθεί ιδιαίτερα από πολλού Γερμανού συναδέλφου μας. Τρίτο σημείο που ανέφεραν και πάλι οι Γερμανοί και οι Πολωνοί συνάδελφοι στην, από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν το θέμα της φορολογίας, δηλαδή η ανάγκη την οποία σημείζονται ευρέως για πρόοδο όσον αφορά την ε, φορολογική εναρμόνιση. Τακτικά αυτό, μηνιαία δηλαδή, όσον αφορά το σύνολο των φόρων. Όπως επίσης αναφέρθηκε και η ανάγκη για πρόοδο για μια ευρωπαϊκή φορολόγηση των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ένα άλλο τέταρτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω αναφέρθηκε από τον Βέλγο συμπρόεδρό μας, δηλαδή οι διεθνεί οργανισμοί αξιολόγηση, Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης και κατά πόσο θα μπορούσε ένας τέτοιος οργανισμός να παρενέβει όταν έχουμε να αξιολογήσουμε το εθνικό χρέος των χωρών μελών. Πέμπτο σημείο και τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι η ισορροπία συνολική μεταξύ της σκέψης για την οικονομική, οικονομική διακυβέρνηση σε σχέση και σε αρμονία με τις πρώτες σκέψεις που αναφέρατε στην προηγούμενη ομάδα δηλαδή για να δούμε κατά πόσο οι συνθήκε αυτής της οικονομικής διακυβέρνηση θα έπρεπε να αποτρέπουν την χρηματοδότηση των ε, μελλοντικών επενδύσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφερε ένας ε, Γερμανός συνάδελφο, το οποίο νομίζω θα πρέπει να επενθυμίσουμε εδώ. Πάντως, γενικά, πιστεύουμε ότι τα μέτρα για την χειραγώγηση, μάλλον για την ε, για τον έλεγχο του εθνικού χρέους δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τις μελλοντικέ επενδύσεις και ένας Ιταλός συνάδελφος μάλιστα αναφέρθηκε στην έκδοση ομολόγων ευρωπαϊκών για την χρηματοδότηση απαραίτητων χρηματοδοτήσεων στην ε, υποδομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος να αναφέρω την ησυχία πολλών συναδέλφων ότι το σύνολο το μέτρων αυτό θα πρέπει βεβαίως να οδηγήσει και στην, στην δημιουργία απασχόλησης και στον στόχο που έχουμε τη καταπολέμησης της ένδυα, τη στόχια. Αυτά, Πρόεδρε, για τη δική μα ομάδα εργασία. Ακούστηκαν πολλά θέματα προς συζήτηση και βεβαίω υπήρξε βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση εάν το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν συνεργαστούν ο καθένα στον τομέα αρμοδιοτήτων βεβαίω, αλλά ακολουθώντα μια κοινή στρατηγική που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή μάλιστα που συζητείται το θέμα του πολέμου των νομισμάτων να προχωρήσει ώστε να είναι ε, ισχυρή και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρεβάνς. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπερές. Θα περάσουμε αμέσως στην έκθεση της τρεις ομάδας εργασίας με θέμα το πώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά στην Ευρώπη. Το λόγο έχει ο κ. Ζόρδι Βλαζοάνα γερουσιαστής από την Ισπανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή, ε, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, κύριοι Στην τρίτη ομάδα εργασία χθε, όπου είχα την τιμή να συμμετάσχω ως εισηγητής, συζητήθηκε η ανάλυση των προκλήσεων που παρουσιάζει η νέα αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο αποτελεί ένας από τους βασικούς πυλώνες της. Οι απόψεις που ακούστηκαν στην τρίτη ομάδα εργασία επιβεβαιώνουν τις απόψεις, τις θέσεις της έκθεσης Μόντι, σύμφωνα με την οποία η γενή αγορά δημιουργεί προσδοκίες και ανησυχίες που σχετίζονται με την πραγματικότητα της κάθε χώρας μέλους και σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η πραγματικότητα ανταποκρίνεται βεβαίως ή αντιστοιχεί σε μια κρίση ενώ σε, ενώ σε άλλες χώρες έχουμε ήδη μια οικονομική ανάκαμψη. Εξάλλου στη συζήτηση αναφέρθηκαν και διάφορες ιδεολογίες όσον αφορά την οικονομική πολιτική που πηγαίνουν από τον καθαρό οικονομικό φιλελευθερισμό με μια υπεράσπιση της οικονομίας αγοράς με κοινωνικές τάσεις. Παρά αυτές τις διαφορές, η πλειοψηφία των ομιλητών αναφέρθηκε στην ανάγκη για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νέας αγοράς που θα έχει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών. Ακούστηκαν διάφορε απόψεις σχετικά με τα υπέρ και τα κατά του ανοίγματο της ενιαίας αγορά και παρόλο που υπήρξαν απόψεις υπέρ του προστατευτισμού και της επιστροφής στον οικονομικό αθνικισμό η πλειοψηφία των παρεμβάσεων κατέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης των ελευθεριών που προϋποθέτει η αγορά. Μεταξύ των μέτρων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν υπό την έννοια αυτή ξεχωρίζουν κάποιες όπως η ενοποίηση των νομοθεσιών των χωρών μελών η μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών και ευελιξία τους και ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής τους. Υπό την έννοια αυτή αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας για, τους, ε, για τις δημόσιες προσλήψεις παρόλο, κάτι που παρόλο που αφορά την ενιαία αγορά επιφέρει σημαντικές ε, γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης αναφέρθηκαν οι ελπίδες και οι επιφυλάξεις σε σχέση με την ε, μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες και ε, ό,τι αυτή εκπροσωπεί. Επίσης συζητήθηκαν άλλα θέματα όπως η καταλληλότητα προώθησης του σήματος Ευρώπη και το στοίχημα για την ε, καινοτομία ως μορφή ανταγωνισμού με τρίτες χώρες. Η αγορά θα πρέπει να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αποφευχθεί μια ρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία θα αποτρέπει τις, ε, από τις χώρες της Ευρώπης να ανταγωνιστούν ε, ισότιμα τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις οι οποίες τους στους διάφορους τομείς, ο, λειτουργούν στους διάφορους τομείς. Αναφέρθηκε επίσης και η απαραίτητη φορολογική εναρμόνιση η οποία θα πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών θα μπορούσε μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να βλάψει την ανταγωνιστικότητα την ευρωπαϊκή. Η ομάδα εργασίας επίσης θεώρησε επιτυχία την συνολική προσέγγιση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ρυθμίσει την ενιαία αγορά μέσω του πακέτου μέτρων που παρουσιάστηκαν ε, τον Οκτώβριο του 2010 ο που παρουσίασε ο κ. Μπαρνιέ, ο αρμόδιος επίτροπος. Η συζήτηση που έγινε στην τρίτη ομάδα εργασίας θα μπορούσε δηλαδή να θεωρηθεί ως καρποφόρα στο μέτρο που οι ομιλίες, οι παρεμβάσεις και οι απόψεις ήταν πάρα πολλές και ποικίλε και έγινε σαφής η σχέση των βουλευτών που έλαβαν το λόγο με την οικονομική πραγματικότητα που επικρατεί στην κάθε χώρα μέλη. Καταλήξαμε στα συμπεράσματα τα οποία αντανακλούν βεβαίω τι διαφορέ απόψει στην ομάδα εργασία και ελπίζουμε να αποτελούσουν ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο, χωρί βεβαίω να αποκλείσουμε άλλε απόψει οι οποίε θα ακουστούν στην διάρκεια τη υπόλοιπη συνεδρίασή μα. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Ζόρδη. Επομένως, ε, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τους τρεις εισηγητές από τις τρεις ομάδες εργασίας. Θα τις έχουμε και γραπτό στις παρεμβάσεις αυτές και θα σας τις διανύμουμε. Είναι κείμενα εξαιρετικά ενδιαφέροντα κατά την άποψή μου και οι ιδέες αυτές είναι χρήσιμες, θα μας εμπνεύσουν στο έργο μας. Στη συνέχεια. Περνούμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο. Από ό,τι έμαθα, ο κύριος Ιβλε Τέχν, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρωθυπουργός του Βελγίου, θα φτάσει στις 10.30. Επομένως θα πάρει το λόγο τότε. Γι' αυτό και ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αλλάξουμε ε, τη σειρά των παρεμβαίνοντων. Και βεβαίως ο, ο πρόεδρος Μπαρόσο είναι πάντοτε εξαιρετικά ευέλικτος και απάντησε θετικά. Θα πάρει εκείνος πρώτα το λόγο και στη συνέχεια ο κύριος Λετέο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι πολύ σημαντικές οι στιγμές αυτές όπου μπορώ να πάρω το λόγο μπροστά σε εκπροσώπους όλων των κοινοβουλίων. Το θέμα δεν είναι θέμα τύπου η ευγενία. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το οποίο θα ήθελα να στείλω. Η πρόκληση σήμερα είναι τόσο δύσκολη που απαιτείται η προσπάθεια όλων. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση και δεν πρόκειται να πετύχουμε αν δεν συνδυάσουμε τη δράση μας σε ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη-μέλη. Απαιτείται ένα κοινό όραμα για να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να πείσουμε τους Ευρωπαίους να συνεργαστούν με τον στόχο αυτό, για τον στόχο αυτό. Η κοινοβουλευτική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Έχετε την δημοκρατική αναγνώριση που απαιτείται και έχετε την δυνατότητα τα μηνύματα αυτά να τα περάσετε σε όλη την Ένωση. Συστηματικά λοιπόν προσπαθώ να ενισχύσω τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διεύρυνση και ευάθυνση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να εντατικοποιήσω τις επαφές τις οποίες έχουμε τώρα κάτω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση να μιλήσουμε μεταξύ μας πολύ, να ακούσουμε ένα τον άλλον ακόμα περισσότερο. Και έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή με μια κοινή θέση. Ένα μήνυμα από την κρίση είναι ξεκάθαρο. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν, οι ιδιαιτέρως ανησυχούν. Ανησυχούν κυρίως για τις θέσεις εργασίας τους, τη δυνατότητα να κρατήσουν τη θέση τους αυτοί που την έχουν, να ξαναβρούν αυτοί που την έχασαν ή να έχουν στο μέλλον αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να σπουδάζουν σήμερα. Ανησυχούν για την εκπαίδευσή τους, την συντάξη τους, την ποιότητα ζωής τους, το περιβάλλον τους και περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαντήσεις. Πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη. Η κρίση αυτή ε, θα έλεγα δημιουργεί ε, συστήματα ελέγχου για τις ικανότητές μας και για την αλληλεγγύη την οποία θα πρέπει να επιδείξουμε ο ένας προς τον άλλο. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο της οικονομικής ανάκαμψης. Υπάρχουν κάποια πρώτα δείγματα βελτίωσης. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα αναπτυχθεί περισσότερο εφέτος από όσο υπολογίζαμε αλλά η ανάκαμψη δεν είναι ακόμα σταθερή και η κατάσταση διαφέρει ιδιαίτερα από χώρα σε χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ για ε, θα έλεγα αδράνεια ε, χώρος. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για κοινή λύση. Η οικονομική πολιτική της Ένωσης έχει μετασχηματιστεί από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε περάσει σε μια βαθιά αλλαγή μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία του αύριο μέσω της στρατηγικής του 2020 για φόρο σταθερή ανάπτυξη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν εξετάσει όλες τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του χρηματοδοτικού συστήματος. Νέα μέτρα έχουν ληφθεί στον τομέα της εποπτείας, σαν παράδειγμα. Αλλά είναι ακόμα υποσυζήτηση. Και κάποια ακόμα δεν έχουν προταθεί. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω ότι θα έχουμε συντελέσει μια επανάσταση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και έχουμε βάλει τα θεμέλια για το μέλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία της μελλοντικής μας οικονομίας είναι να εφαρμόσουμε τα προγράμματα τα οποία δεν θα έχουν προηγούμενο θα έλεγα στο μέγεθός τους και στο εύρος τους. Βέβαια πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα οι συνέπειε της κρίση φέτο είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Εξέθεσε θα έλεγα πως δεν καταφέραμε να συγχρονιστούμε με τις προκλήσεις οι οποίες μας περιβάλλουν και έτσι τα θεμέλια μας κλονίστηκαν. Τον Μάιο θα εφαρμόσουμε το νέο μηχανισμό σταθεροποίησης και το Σεπτέμβριο προτάθηκαν νέες, ε, έγιναν νέες προτάσεις για τον τομέα της εποπτείας ε, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συναλλαγών. Όλα αυτά ε, είχαν φυσικά σαν προαπέτηση να υπάρξει μια ισχυρή συνένεση η οποία υπήρξε μετά από πολλαπλές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τον προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τις απόψεις αυτές και πρότεινε την δημιουργία ενός συνολικότερου μηχανισμού αντιμετώπιση της κρίσης. Τις προτάσεις αυτές τις εξετάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με έντονο επεμβατικό τρόπο. Απαιτείται η υποστήριξή σας γιατί θα προσδώσετε περαιτέρω νομική ασφάλεια και βεβαιότητα στον μηχανισμό τον οποίο χρειάζονται οι περισσότερες χώρες. Οι μελλοντικές αλλαγές δεν θα είναι τόσο μεγάλου μεγέθους, δεν θα χρειαστεί να είναι τόσο μεγάλου μεγέθους, δεν θα αλλάξουν οι αρμοδιότητες, θα έλεγα, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόβλεψη ε, νομίζω είναι το σύστημα αυτό να λειτουργήσει από 2013 όπου ο προσωρινός παρόν μηχανισμός που ισχύει θα τερματιστεί. Νομίζω ότι έτσι θα βάλουμε τα θωστά θεμέλια για το μέλλον. Αλλά αυτές οι προσπάθειες σταθερότητας δεν είναι αφέ αυτές, θα έλεγα, η πανάκια. Απαιτούνται περισσότερα μέτρα. Πρέπει να κάνουμε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Και αυτό ακριβώς είναι η στρατηγική μας η καινούργια την οποία προτείνουμε, η στρατηγική 2020. Προσβλέπουμε στο μέλλον, σε ένα μέλλον έξυπνο, σε ένα μέλλον ευφυές, σε ένα μέλλον αηφόρο πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Θα τις πετύχουμε τις αλλαγές αυτές μόνο από κοινού. Και φυσικά τα κοινοβούλια εδώ καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και το ευρωπαϊκό και τα υπόλοιπα. Απαιτείται λοιπόν η υποστήριξή σας για να αποδείξουμε, να προωθήσουμε, να εξηγήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα, θα πρέπει να προλάβουμε θα έλεγα την κατάσταση με τις πρώτες προτάσεις μας. Ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο λοιπόν που θα οδηγήσει σε έναν μηχανισμό που θα καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, θα βασιστεί στην εσωτερική αγορά, θα προωθήσει την αηφορία, θα προωθήσει την καινοτομία, θα καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ευέλικτη Αυτές οι ευέλικτες πρωτοβουλίες και η ψηφιακή ατζέντα την οποία έχουμε ξεκινήσει υπογραμμίζει θα έλεγα τον ρόλο που παίζει το διαδίκτυο έτσι ώστε να έρθουμε στην ίδια ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων με τους ανταγωνιστές μας. Η καινοτομία θα πρέπει να συνεχιστεί και στον τομέα της έρευνας και στον τομέα της επιστήμης έτσι ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και της προσπάθειας επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα καταπολεμήσουμε και την ένδια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα βελτιώσουμε τα μέτρα υποστήριξης της νεότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα είναι μια κοινή, θα έλεγα, πηξίδα για την πορεία μας στο μέλλον. Για να το πετύχουμε όμως χρειαζόμαστε και νέα μέσα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του παρελθόντος που πολλές φορές δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Γι' αυτό τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν τα προγράμματα αυτά περιοριστούν σε αγραφειοκρατικές προσπάθειες τότε θα χάσουμε πολύ χρόνο. Αν πετύχουν όμως τα προγράμματα αυτά να συνδυάσουν τις εθνικές οικονομικές πολιτικές με την ουσία της ευρωπαϊκής διάστασης θα είναι οι μοχλοί οι οποίοι θα προκαλέσουν τις αλλαγές που απαιτούνται για την οικονομική μας ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν από το πρώτο στάδιο να συνεργαστούμε με τα κοινοβούλια έτσι ώστε να υπάρξει σωστή ενημέρωση και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Όσο πιο δύσκολες είναι οι μεταρρυθμίσεις, τόσο περισσότερο απαιτείται μια συνένεση ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν ολοκληρωθούν τα προγράμματα αυτά, προφανώς δεν θα έχει τελειώσει η προσπάθεια. Οι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά, να δούνε τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει τόσο καλά και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και να ελέγξουν δημοκρατικά τις κατευθύνσεις της οικονομίας μας. Γνωρίζω ότι ορισμένα εθνικά κοινοβούλια ανησυχούν για τις πιθανές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δημοσιονομικέ στις δημοσιονομικές τους ε, ε, αρμοδιότητες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μας αυτή. Ελπίζω όλες αυτές τις ανησυχίες να τις αποσύρουμε. Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική για το συνδυασμό των εθνικών προσπαθειών. Σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών και όσο περισσότερες πληροφορίε έχουμε τόσο πιο ενισχυμένη θέση θα έχουμε στο παιχνίδι αυτό. Σωστές πληροφορίε για τις μακροοικονομικές τάσεις, για τη φορολογική κατάσταση και για τις προσπάθειες μεταρρύθμισης. Έτσι θα αλλάξουμε τα πράγματα. Η κρίση μας έδειξε ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι οι ε, αποφάσεις σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η οικονομική πολιτική λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αυστηρά σαν εθνικό φαινόμενο. Αυτό είναι προφανές και όποιος αρνείται αυτό το γεγονός αρνείται την πραγματικότητα. Η αλληλεξάρτηση είναι εκεί, ακόμα και παγκόσμια θα έλεγα αλληλεξάρτηση. Πώς μπορούμε εμείς να υποστηρίζουμε την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και να αρνούμεθα τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς πιστεύουμε ότι απαιτείται μια συνεκτική και συγκριτική αντιμετώπιση για να δουλέψει το σύστημα αυτό. Να υπάρξουν ξεκάθαρα στάνταρτς επίπεδα για τα φορολογικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο όπως επίσης και για τα δημοσιονομικά μέτρα και αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να συμβαδίζουν φυσικά με τον δημοκρατικό έλεγχο και με μια στενότερη εμπλοκή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμίζω, δημοκρατικά άμεσα εκλέγεται, έχει πλήρη νομιμοποίηση, δεν είναι κοινοβούλιο δευτέρας κατηγορίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, ιδιαίτερα μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί σε εθνικό επίπεδο κάποιοι πολιτικοί από τις εθνικές πολιτικές τάξεις δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών οργάνων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συντονίσουμε τα πράγματα για να απαντήσουμε στην κρίση, αλλά δεν θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία κάναμε στο παρελθόν. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία, μια οικονομία η οποία θα είναι αυτή που απαιτείται να είναι μια οικονομία που να βασίζεται σε βασικές αρχές. Μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το λέγει αυτό και η συνθήκη της Λισαβόνας. Μια οικονομία που να αναγνωρίζει τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στα έφτραστα σώματα, στρώματα των κοινωνιών μας. Και μια οικονομία επίσης με περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων διοξιδίου του άνθρακα στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει εμείς να μην εγκαταλείψουμε τις αξίες μας όμως γι' αυτό, πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, πρέπει να σεβαστούμε την κοινωνική διάσταση της προσπάθειας μας και αυτό θα γίνει με συνδυασμό της εθνικής διάστασης με την ευρωπαϊκή διάσταση. Συνεπώς λοιπόν σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα συνεργαστώ όσο καλύτερα μπορώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε και φίλε. Δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Λετέρμα. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να δείξουμε ε, την ευελιξία που έχουμε τόσο εμείς όσο και το Βέλγιο. Γι' αυτό λοιπόν να ξεκινήσουμε ήδη τη συζήτηση με τους συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ημιλητών και όταν έλθει ο κύριος Λετέρμα θα διακόψουμε για να ακούσουμε την ομιλία του. Να σας υπενθυμίσω τη διαδικασία. Κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του τρία λεπτά. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα και να μην ξεπεράσετε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Χθες λειτουργήσαμε με τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας. Δηλαδή, δεν είστε υποχρεωμένοι να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά βεβαίως μπορείτε Όταν τελειώνει ένας ομιλητής, εάν μπορεί, κάποιος άλλος ομιλητής μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να κρατάει τη γαλάζια τα ε, κάρτα. Επομένως, θα ρωτηθεί, θέλει να δεχθεί την ε, ερώτηση του άλλου συναδέλφου. Εάν ναι, τότε έχει 30 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα για να ε, κάνει το ερώτημά του, να χρησιμοποιήσει δηλαδή τη γαλάζια κάρτα και έχει άλλα 30 δευτερόλεπτα ο ερωτώμενος να απαντήσει. Δύο φορές μπορεί ένας συνάδελφος να χρησιμοποιήσει τη γαλάζια κάρτα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν για μένα τώρα που δίνω την προεδρία της συνεδρίασης στον συνάδελφο κύριο Ντεμάγερς, αντιπρόεδρο της Γερουσίας του Βελγίου και δήμαρχο της πόλης της Λιέγης. Το οποίο είναι βέβαια προνόμιο. Θα συμφωνήσετε όλοι όσοι έχετε επισκεφθεί τη Λιέγη. Και θα έρθω εγώ να καθίσω δίπλα στο φίλο μου τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να προεδρεύσω αυτής ε, της τόσο εξέχουσα συνέλευσης. Να δώσω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο στην κυρία το Βίσαιτε από τη Λιθουανία. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλωσορίζουμε την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την υλοποίηση όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων μετά την σοβαρή κρίση που έπληξε την Ευρώπη και κυρίως το χρηματοπιστωτικό τομέα. Έδειξε η κρίση ξεκάθαρα την αναγκαιότητα για συνολικές και γενικές ρυθμίσεις Θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν ξέρω όμως άμα θα έχει αποτελέσματα αν θεσπιστεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι χρηματαγορές, ξέρετε, είναι παγκόσμιες. Επομένως, η Ευρώπη ως πολύ σημαντικός παίκτη οικονομικός στο διεθνές στερέωμα θα πρέπει να ασκήσει πίεση, πίεση για έναν παγκόσμιο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι τράπεζες δημιούργησαν την κρίση και μάλιστα αυτές είναι αυτές που ωφελούνται και περισσότερο από την κρίση σήμερα. Γίνεται λόγος για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ξέρετε ε, πόσο υψηλό είναι το χρέος των κρατών μελών. Οι τράπεζες ε, αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες, ουσιαστικά βγάζουν κέρδος από το υψηλό χρέος των κρατών μελών, χωρίς ε, να μετακυλίουν ε, αυτά τα κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ συχνά έχει δοθεί, έχει δοθεί υπερβολική βοήθεια στις τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για τις τράπεζες και να τις εξαναγκάσουμε να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ως προς τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, καλό θα ήταν να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να καλέσω τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να μην μένουν μόνο σε δηλώσεις περί αλληλεγγύης, αλλά να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις και κυρίως στο θέμα της ενέργειας. Πολύ συχνά στα ενεργειακά θέματα βλέπουμε ότι το διμερές επίπεδο είναι πιο σημαντικό. Χαίρομαι διότι βλέπω ότι εμπιστεύεστε τα εθνικά κοινοβούλια. Η ανταλλαγή πληροφοριών περί δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αρμοδιότητα, έχουν μέσα και εργαλεία για να ασκούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των κυβερνήσεων, κυρίως σε θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω διότι ε, έχετε μείνει εντός του χρόνου που σας είχε δοθεί στρέφουμε προς τον δεύτερο μιλητή, τον κύριο Αντρέη Καλαζεύσκη από την Πολωνία. Έχετε το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η καλύτερη, χρημα... η καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη είναι μια ανάγκη στην Ευρώπη ως απάντηση για την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τις ε, συνθήκες που δημιούργησαν την ανάγκη αυτή, ώστε να έχουμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών και να έχουμε ένα πλαίσιο διαχείρισης των οικονομικών ε, κρίσεων. Αυτή είναι στόχη η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι απειλές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως στρατηγικά θα πρέπει να αυξήσουμε, να μεγαλώσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την νέα αγορά 10 χρόνια μετά από την έναρξη αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι η ανταγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντίστοιχα ανάλογη με την ανταγωνιστική θέση των χωρών μελών και οι χώρες αυτές βεβαίως ανταγωνίζονται και μεταξύ τους υπάρχει εσωτερικό ανταγωνισμό και αυτό ο εσωτερικό αγωνισμό είναι μια προστιθέμενη αξία. Όμω, τη χθεσινή τη συζήτηση, σχετικά δηλαδή με το θέμα της, ε, του εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ των, δηλαδή, χωρών μελών και το θέμα των ε, συστήματων φορολογίας ε, είχαμε κάποιες αρνητικές απόψεις. Δηλαδή είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο ή όχι όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Συζητήσαμε λοιπόν και τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την φορολογία ώστε να χρησιμοποιούμε όλη την ίδια γλώσσα. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά όσον αφορά το συντελεστή φορολόγησης και το κόστος το εργατικό, ο ανταγωνισμός ο αυτός θα παραμένει. Ο κύριος Μπαρόζο μίλησε για νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται με νέες επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε επενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΙΠΑ, ε, Ινδία, Βραζιλία, τρίτες χώρες γενικότερα και να τους δώσουμε κίνητρα να επενδύσουν. Και για να δοθούν αυτά τα κίνητρα για να επενδύσουν θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως μια ρύθμιση του εσωτερικού ανταγωνισμού που αφορά τη φορολογία, το εργατικό κόστος, ε, την παροχή ε, δανείων, όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας προτείνω να περάσουμε στην τρίτη ομιλία. Ο κύριος Χάρμπορ, Ευρωβουλευτής, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ως Πρόεδρος στην ε, Επιτροπή για την Ιάγορα στην ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέδρευσα χθε και συζητήσαμε πολλά θέματα αλλά κυρίως το πώς θα μπορούσε να οκληρωθεί η νέα αγορά. Θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την εργασία που έχει κάνει η δική μου επιτροπή. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στην στρατηγική 2020. Όπως ξέρουμε τώρα, πριν δύο εβδομάδες δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει την ε, ε, το νόμο την πράξη για την νέα αγορά μετά από διαβουλεύσεις και πολλές προτάσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Σημείωσα ότι ο πρώτος της Επιτροπής αναφέρθηκε για την ύπαρξη δανείων. Ξέρω βέβαια ότι δεν αναφέρθηκε σε αυτή την ε, πράξη νέας αγοράς, αλλά φαντάζομαι θα το αναφέρει αργότερα, επειδή ακριβώς αυτή η ιδέα ήταν της Επιτροπής μου και ακριβώς δείχνει το τι μπορούμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο και λέμε στην Κομισιόν ότι δεν θεωρούμε ότι η στρατηγική 2020 ότι έχει το αρκετό ύψος για να πετύχει τους στόχους και ε, τα, τα απαραίτητα στοιχεία για να βγει η Ευρώπη από την κρίση. Γι' αυτό ακριβώς λέμε στην ε, Κομισιόν ότι το θέμα των, διεθνών των δημοσίων διαγωνισμών δεν λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε γραφειοκρατία. Μάλλον έχουμε γραφειοκρατία αντί να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθά τι επενδύσει. Και πάλι νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προτεραιότητα έχει παραβλεφθεί. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πώ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να περάσουμε στην κατάλληλη στρατηγική. Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο σημείο που θέλω να σα αναφέρω εδώ στου συναδέλφου και ε, με την παρουσία τη Κομισιόν και είναι το εξή. Αν τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να διαδραματίσουν τον απαραίτητο και ουσιώδη ρόλο τους σε συνεργασία με εμά, ώστε να τονίσουμε τη σημασία της ενιαίας αγοράς και σε σχέση πάντοτε με τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες Ευρωπαίους θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ παραπέρα όσον αφορά τις στρατηγικές πολιτικές μας. νομίζω ότι δεν είναι και τόσο χρήσιμο να μας στέλνει η Κομισιόν μεγάλο αριθμό προτάσεων για τις οποίες είμαστε ελάχιστα προετοιμασμένοι με ελάχιστη προθεσμία λίγων εβδομάδων να απαντήσουμε. Αυτό δεν μας βοηθάει. Αυτό που θα πρέπει να μας επιτρέψει, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει μάλλον να συμμετάσχουμε στις μελλοντικέ ε, προτάσεις και στρατηγικές είναι ο εξή. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα και θα το κάνω ταχύτατα για να μην ξεπεράσω τον χρόνο, Πρόεδρε. Για την αμοιβή αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων, ξέρουμε ότι η Κομισιόν θα θεσπίσει μια αναθεώρηση Μελλοντικά, το 2011, εμείς θα εκπονήσουμε μια σημαντική στρατική μελέτη για αυτό το θέμα και υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ήδη είχαν επαφές με εθνικούς βουλευτές για να σας μεταφέρουν τις ανησυχίες μας για την πρόταση αυτή και διάφοροι από εσάς είχατε συμμετάσχει σε αυτές τις συναντήσεις. Τώρα, συναδελφοί πρόεδροι τη Επιτροπή. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση, δηλαδή θα πρέπει να έρθετε εσεί στην Επιτροπή σαν τη δική μου και να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε τι προτάσει τη ε, Κομισιόν. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και εσεί, Πρόεδρε, ελπίζω ως διαχειριστής των διακοινοβουλευτικών σχέσεων νομίζω ότι θα πρέπει οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν την κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε να έχουμε δώσει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να προτείνω τώρα στον τέταρτο μιλητή να πάρει το λόγο. Ρόμπερτ Λούγκορ. Από την Ομοσπονδιακή Βουλή της Αυστρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τράπεζες παίρνουν τεράστιες πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1%. Και τι κάνουν τα χρήματα αυτά, δεν εκτίθενται σε κανένα κίνδυνο και σημειώνουν κέρδη τα οποία από έτος σε έτος αυξάνονται τουλάχιστον κατά 10% χωρίς κανένα κίνδυνο και με την πλήρη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς βλέπουμε ότι από αυτή την κρίση αυτοί οι οποίοι κέρδισαν, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι οι τράπεζες λόγω του χαμηλού ευρωπαϊκού επιτοκίου, το οποίο δεν ωφελεί αυτούς που θα έπρεπε να ωφελήσει, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όχι μόνο στη δική μου χώρα, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρώπης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις απασχόλησης αυτές όταν πρέπει να δανείζονται ε, πρέπει να δανείζονται μέχρι και με 7% γιατί κανένας δεν καλύπτει με εγγυήσει ε, τα χρήματα τα οποία παίρνουν. αυτό το χαμηλό επιτόκιο με το οποίο δανείζει χρήματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυστυχώς δεν επιτρέπει να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας όπως αυτό είχε προβλεφθεί, όπως αυτή ήταν η λογική αν θέλετε. Και δυστυχώς κάποιοι ωφελούνται από την κατάσταση αυτή αλλά ωφελούνται με τέτοιο τρόπο που κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί μια νέα κρίση και δεν θα τονωθεί η οικονομία και δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. μέσα σε 10-15 χρόνια θα ζούμε μια κατάσταση εντελώ διαφορετική από τη σημερινή. Σήμερα έχουμε υψηλά επίπεδα εργατικού δυναμικού αλλά λίγα παιδιά και σε 10 χρόνια θα έχουμε το αντίθετο πρόβλημα. Θα υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού για δημογραφικούς λόγους. Τι σημαίνει αυτό βέβαια, πρέπει να κάνουμε περισσότερα παιδιά σήμερα ή μήπως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο της μετανάστευσης. Μια μετανάστευση με ποιοτικά κριτήρια, μια μετανάστευση επιλεκτική, μια μετανάστευση η οποία θα επιτρέπει τον ερχομό στην Ευρώπη αυτών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και αρμοδιότητες για να καλύψουν τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που θα έχουμε ανάγκη του χρόνου. Έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες στις χώρες μας που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα επίπεδα θα έλεγα εμπειρογνωμοσύνης και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Απαιτούνται λοιπόν νέες ρυθμίσεις ιδιαίτερα σε σχέση με τον κανονισμό για τη χορήγηση ασύλου. Ε, αυτή την εποχή σημειώνεται μια τεράστια εισρωή ε, μεταναστών ή παρανόμων εν πάση περιπτώσει μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σας ευχαριστώ. Νομίζω θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, πέμπτη ομιλήτρια, την κυρία Ολέσοσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Οι προκλήσεις τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πέρα από την οικονομική κρίση έχουν δημιουργηθεί νέα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και θα συζητήθηκαν βέβαια και στα πλαίσια των ομάδων εργασίας. Απασχόληση, οικονομική διακυβέρνηση, δημιουργία ενιαίας αγοράς, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία χρήζουν συζήτησης και απάντησης. Νομίζω ότι αν δώσουμε τις σωστές απαντήσεις θα έχουμε νέες δυνατότητες ε, ανάπτυξης της οικονομίας μας. Εγώ είμαι μέλος της Οικονομικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Πολωνικής Βουλής. Και ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι δημόσιες προμήθειες. Οι νομικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κρατικές προμήθειες είναι μερικές φορές ε, δυνατόν να γίνουν σεβαστές από τον επιχειρηματικό κόσμο. Αλλά σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις και όπου υπάρχουν ευκαιρίες για α, δημόσιες προμήθειες, οι επιχειρηματίες δεν είναι πολλές φορές εύκολο να πάρουν μέρος στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, γιατί είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και διαμαρτύρονται έντονα για τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Βέβαια και αυτοί έχουν ευθύνε για την πλήρη τήρηση των μέτρων, γιατί τα μέτρα αυτά είναι μερικές φορές απαραίτητα για την επιτυχή κατάληξη αυτών των διαδικασιών προμήθειας. γιατί λογικό είναι να επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν τις περισσότερες εγγυήσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν να καταρτίζουν σωστά τον επιχειρηματικό κόσμο έτσι ώστε να γνωρίζει τι κινδύνους αντιμετωπίζει συμμετέχοντας σε τέτοιες διαδικασίες διαγωνισμούς ε, που οργανώνει το δημόσιο και να τους προετοιμάζει σωστά για την επιτυχή προσφορά τους. Πολλά κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες κατάρτισης των επιχειρηματικού, του επιχειρηματικού κόσμου για να γνωστοποιήσουν και στο ευρύτερο κοινό τι ακριβώς συμβαίνει, τι νέες καινοτόμες ιδέες μπορούν να βρεθούν, έτσι ώστε να αναζητήσει ο επιχειρηματικός κόσμος νέους επενδυτικούς χώρους και να κάνει προτάσεις οι οποίες να είναι φιλικές για την οικονομία και το μέλλον μας. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιους τομείς μπορούν οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους και σε ποιους τομείς τα κράτη μπορούν να ωφεληθούν από τις σωστότερες αυτές συμπεριφορές έτσι ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα ναι να είναι περισσότερο κερδοφόρα αλλά να μην δημιουργεί κινδύνους. Το θέμα δεν είναι μόνο να ξεκινήσουμε νέες επιχειρήσεις. Στη δική μου χώρα καταφέραμε το πρόβλημα των νέων επιχειρήσεων να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χίλτα Φιγκερέιδο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση να έχουμε τα εξής υπόψη μας. Καταρχάς, η ανεργία καλπάζει, η ανισότητα καλπάζει και η φτώχεια οξύνεται. Έχουν τονιστεί όλα αυτά, αλλά έχει υποθεί επίσης ότι την κρίση την προκάλεσαν οι τράπεζες καταρχάς, ενώ από την άλλη οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες υποφελούνται από την κρίση σήμερα. Κατά δεύτερο λόγο. Και γι' αυτό έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλα αυτά τα προβλήματα στη χρηματοδότησή τους. Ε, και η κατάσταση επιδεινώνεται με τα διάφορα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόζονται στις χώρες που αντιμετωπίζουν και τα πιο μεγάλα προβλήματα. Χώρες ε, ασθενείς ως προς τα οικονομικά τους. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα λιτότητες εφαρμόζονται αυστηρά βάσει των εντελώς παράλογων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και η κατάσταση έτσι γίνεται χειρότερα. Χειρότερη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα ή στην Ιρλανδία, αναφέρομαι και στην Πορτογαλία, όπου αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δραματική. Στο, μέλλον, με τέτοιου είδου παράλογα μέτρα θα έχουμε περισσότερη ανεργία, περισσότερη φτώχεια, περισσότερες ανισότητες και ασυμμετρίες. Με άλλα λόγια, και φτάνω εδώ στο, στη δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Η κρίση ουσιαστικά δημιουργεί ακόμα λιγότερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώνει τη φτώχεια σήμερα που υποτίθεται ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Εάν δείτε τα στοιχεία, τα αριθμητικά, στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στη φτώχεια θα διαβάσετε ότι έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πώς μπορεί να γίνει αντιληπτή αυτή η κατάσταση. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλά για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ταυτοχρόνως επιβάλλει μέτρα και κανόνες για να τηρούνται τα διάφορα σύμφωνα σταθερότητας μέτρα και κανόνες οι οποίοι οξύνουν το επίπεδο της φτώχειας. Και η τρίτη μου παρατήρηση είναι η εξής. Είναι ζωτική σημασία να μην είναι η χρηματοπιστωτική και οικονομική βιωσιμότητα βασικό μας μέλημα. Βασικό μας μέλημα πρέπει να είναι η κοινωνική βιωσιμότητα ή τουλάχιστον να εξισορροπηθούν αυτά τα δύο. Ας μην συνεχίσουμε με αυτές τις ε, κοντόφθαλμες πολιτικές που επιδεινώνουν τις ε, κοινωνικές εντάσεις και που εξασθενούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και εξασθενούν τη συνοχή του, εάν υπάρχει αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον των παιδιών μας, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ιβ Λετέρμ, όχι, με συγχωρείτε. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα έρθει ο κύριος Λετέρ. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ιβλετέρ. Με καθυστέρησε λόγω της ε, ε, μιας τελετής στην οποία έπρεπε να παρουσιαστεί. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως ανακάστηκα να παραστώ στην εκκρεώσιμο ακολουθία του κυρίου Ντουκένε και γι' αυτό καθυστέρησα, θα γίνει σήμερα και θα πρέπει να φύγω. Σήμερα το πρωί ήμουν σε συνεδρίαση του Υπουργικού Μα Συμβουλίου για το προπολογισμό μας και μπορώ να διαβεβαιώσω τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Μπαρόζο ότι ο προπολογισμό του Βελγίου θα, είναι, ε, θα τηρεί αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν για την καθυστέρηση και ξεκινώ αμέσως λέγοντας ότι είναι ευκαιρία πλέον να μιλήσουμε για την έξοδό μας από την κρίση. Δύο χρόνια μετά, την, μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Ουσιαστικά έτσι δείξαμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσαμε αρκετά γρήγορα θα ήθελα. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλήσω και για τη Βελγική Προεδρία. 52 μέρες έμειναν μέχρι να τελειώσει. Λίγη υπομονή παρακαλώ. Νομίζω ότι ε, καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, ε, σεβαστήκαμε και το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν θέλαμε καθόλου το πρόγραμμά μας να έχει αμυγός βελγική χρειά. Αντιθέτως, προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε θεσμικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θέση του του εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, τα νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών οργάνων και προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε ως διαμεσολαβητές στη Βελγική Προεδρία για να ε, διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και να ολοκληρωθεί η εξέταση όσο δυνατόν περισσότερων φακέλων. Τούτων λεχθέντων. Και θα επανέλθω γιατί στο θέμα αυτό ε, γιατί είναι και το θέμα των συζητήσεών σας. Ως προς την κρίση, ως προς την οικονομική πολιτική, την χρηματοπιστωτική, τη δημοσιονομική κρίση, όλα αυτά ήταν στις προτεραιότητές μας, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η κοινωνική πολιτική, η πολιτική συνοχής, στην οποία δεν είχε δώσει ε, πολύ μεγάλη προσοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική περιβάλλοντος, το κλίμα, οι κλιματολογικές αλλαγές, σύνοδος της ε, Κανκούν και η εξωτερική διάσταση με τη, ως προς τη διεύρυνση. Και σε αυτά εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτά εν ολίγης σε, ήταν τα πέντε χαρακτηριστικά ε, μέληματα της Βελγικής Προεδρίας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να μιλήσω για τις βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εγγύς μέλλον. Δεν θα πρωτοτυπήσω Σίγουρα χρειάζεται καλύτερη οικονομική διαχείριση. Όλα αυτά τα υπογράμμισε το Συμβούλιο στη Σύνοδο της 28 στα τέλη Οκτωβρίου. Επίσης, οι διατάξεις για τον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, η πολιτική για την καινοτομία και την εσωτερική αγορά και η εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας αλλά και της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού η οποία θα ολοκληρωθεί εντός ολίγου. Λοιπόν, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης Οκτωβρίου για το θέμα αυτά. Δώσαμε έμφαση στην ε, μακροοικονομική επιτήρηση ο κύριος Φαν ήταν επικεφαλής των ειδικών ομάδων που κατάρτισαν τις αντίστοιχες εκθέσεις. Έξι προτάσεις ε, είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να ενισχυθεί το σύμφωνο σταθερότητας, να έχουμε διάφορα μέτρα, ενδεχομένως και κυρώσεις. Έγινε συζήτηση για όλα αυτά αλλά και ενδεχομένως για οικονομικές κυρώσεις. Δεν θα επαναλάβω πράγματα που γνωρίζετε ήδη. Το σημαντικό είναι ότι οι κυρώσεις αυτές θα μπορούν να εφαρμόζονται με πιο αυτόματο τρόπο στο μέλλον. Και αυξάνεται η σημασία που έχει το κριτήριο του 60% ως προς το ΑΕΠ και το ε, έλλειμμα. Έγινε συζήτηση και για το επόμενο εξάμεινο από την αρχή του 2011, το ευρωπαϊκό εξάμεινο δηλαδή, να παρουσιάζονται ταυτοχρόνως τα προγράμματα σταθερότητας για κάθε κράτος μέλος, αλλά και τα προγράμματα για εθνικές μεταρρυθμίσεις βάσει αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Φασικές αρχές για ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διαχείριση των κρίσεων, συμφωνήσαμε πάνω σε όλα αυτά βάσει του προτάσεων που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά και ε, με βάση τις κατευθυντήριες ε, γραμμές του ε, συστήματος για την διασφάλιση και την προστασία του ενίου νομίσματος. Επίσης, εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα υιοθετήσαμε συγκεκριμένα κείμενα για τις τέσσερις νέες αρχές που θα εποπτεύουν το χρηματοπιστωτικό τομέα, τον κλάδο των ασφαλίσεων αλλά και τις αγορές και θα υπάρχει και ένα συμβούλιο, το board, που θα έχει τη γενικότερη εποπτεία. Αλλά και θα έχουμε ρυθμίσεις ε, για την διαχείριση εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης. Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί και σε επίπεδο Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί νομοθετική διαδικασία με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε διάφορες φιλοδοξίες για τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο συνάδελφος Reinders μου είπε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά και ότι διαφαίνεται συμφωνία ως προς το θέμα αυτό. Επίσης, η Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Σίγουρα ο κύριος Μπαρόσο ε, σας μίλησε για αυτήν. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Είναι σημαντικό να διδαχθούμε από τις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις της στρατηγικής της Λισαβόνας για να έχουμε ένα πακέτο με μεγαλύτερη συνοχή, ε, με καλύτερη στρατηγική δηλαδή, πιο εύρωστη, με ορίζοντα το 2020. Τώρα, ως προς την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, ε, την κοινωνική ένταξη έχουμε υιοθετήσει στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καθορίσαμε την 12η Νοεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία για να τεθούν στόχοι και σε εθνικό επίπεδο στα διάφορα αυτά πεδία και να προταθούν τα αντίστοιχα μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Έχουμε την ε, πρωτοβου... τις βασικές πρωτοβουλίες όπως είναι η ψηφιακή Ευρώπη και η κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα του Ιουνίου και σε εθνικό επίπεδο η δουλειά που έχει γίνει για τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εισαχθούν σε θεσμικό επίπεδο για να επιτευχθούν οι στόχοι στους πέντε αυτούς βασικούς τομείς. Βεβαίως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 θα έχει νόημα μόνο εάν αξιοποιηθεί για να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση. Η μακροοικονομική στρατηγική, η δημοσιονομική στρατηγική είναι εξίσου σημαντικές ως συνοστώσεις. Είναι συμπληρωματικές αυτές οι τρεις πολιτικές, θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, η μία να στηρίζει την άλλη. Αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση, πιστεύω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τη χαρακτήριζα ως επαναστατική. γιατί βελτιώνουμε ιδιαίτερα την συνεργασία μας στα θέματα αυτά. Το τρίτο στοιχείο είναι η εσωτερική αγορά και η μετανάστευση. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Εδώ έχω και τον διπλωματικό μου σύμβουλο. Προσπαθεί να πείσει ιδιαίτερα τους Ισπανούς συναδέλφους και τους Ιταλούς που συνάντησα την προηγούμενη εβδομάδα για να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα, κύριε Πρόεδρε, σε ένα θέμα που συζητάμε 30 χρόνια, το θέμα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Είναι απαράδεκτο οι βιομηχανίες μας, οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ένα κόστος εννέα φοράς υψηλότερο από ότι οι Αμερικανοί συνάδελφοί τους για να καταθέσουν μια αίτηση για τη χορήγηση ενός τέτοιου διπλώματος. Κάνουμε προσπάθειες και για τη γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κομβικό θέμα, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα και σήμερα το πρωί το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα βέβαιο λόγω των αντιδράσεων κατανοητών ίσως ε, κάποιων ε, συναδέλφων σε άλλες χώρες. Υπάρχει επίσης και το θέμα της ενιαίας πράξης και της ολοκλήρωσης μάλλον της εσωτερικής αγοράς και των εμποδίων τα οποία θα πρέπει να αποσυρθούν. Έχουν εντοπιστεί πλέον και το Συμβούλιο περιμένει ουσιαστικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα πρώτα 50 εμπόδια από τα 150 τα οποία έχουν ανοιχνευθεί στα πλαίσια της πολιτικής για την εσωτερική αγορά και την καινοτομία υπάρχουν μέτρα στα πλαίσια των ελευθέρων συναλλαγών που θα ενισχύσουν την οικονομία μας και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς μας. Ελπίζω ότι τον Σεπτέμβριο ήδη σημειώθηκε μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Κορέα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές ε, στα πλαίσια μιας ευρύτερης σφαιρικού τύπου θα έλεγα συνολικής συμφωνίας κάτι το οποίο είναι μια καινοτομία στα πλαίσια των συνάψεων τέτοιου είδους συμβάσεων. Τέλος, και στα πλαίσια όλων αυτών των πολύ σημαντικών θεμάτων θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα θεσμικά όργανα. Δώσαμε σκληρή μάχη για την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, τώρα τα όργανα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν σύμφωνα με τη νέα συνθήκη. Για μας αυτό είναι μια βασική προτεραιότητα. Ελπίζουμε οι νομοθετικές αυτές προσπάθειες ε, να ολοκληρωθούν σε κάποια φάση. Έχουμε ήδη προωθήσει 20 νομοθετικά κείμενα και τα έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη βδομάδα σαν παράδειγμα ελπίζουμε να κλείσουμε τον προϋπολογισμό του 11 που για πρώτη φορά θα αποφασιστεί επί τη βάση της λεγόμενης στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαλέκτου καθαρής συνεννόησης euh, συναπόφασης σύμφωνα πάντα με τις συζητήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει για το θέμα των ιδίων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να μπορέσουμε αυτή την εβδομάδα να κλείσουμε το θέμα. Η προθεσμία είναι η 15η Νοεμβρίου και οι συναντήσεις έχουν ήδη καθοριστεί για αύριο και μεθαύριο για να δούμε αν πράγματι μπορούμε να καταλήξουμε στα πλαίσια ενός ποσοστού αύξησης των δαπανών περιορισμένου μεν, σεβόμενοι τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ που έχουν όμως εξελιχθεί και που όλο και περισσότερο εδώ εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορέσουμε ελπίζω να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο σας έδωσα τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η Βελγική Προεδρία το οικονομικό κομμάτι, την μεσοπρόθεσμη πολιτική, τη μακροπρόθεσμη πολιτική, το νομοθετικό πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του Συμβουλίου του τέλος Οκτωβρίου, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020, ολοκλήρωση των μέτρων για την οικονομική εποπτεία και ε, θετικό ρόλο για να βελτιωθεί η αξιοπιστία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα, ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ καλύτερα. Και εσείς και ο κύριος Μπαρόσο μπορεί, δεχτήκατε μάλλον να δώσετε και απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα σας τεθούν. Πρέπει να σεβαστούμε τον χρόνο όμως. Πρέπει να δηλώσετε τώρα αν θέλετε να καταθέσετε ερωτήσεις και θα κλείσουμε τον κατάλογο των ερωτήσεων άμεσα. Πρώτη ερώτηση από τον κύριο Γκόραν Πέτερσον από την Σουηδική Βουλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη. Επειδή μόνο μέσω ανάπτυξης μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Διάφοροι ομιλητές τάχθηκαν υπέρ του να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις μέσω του προπολογισμού της Ένωσης. Αυτό είναι σωστό. Όμως, αντί να αυξάνεται ο προπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την διαχείριση του υπάρχοντος προπολογισμού. Δηλαδή, σε αυτόν τον προπολογισμό υπάρχουν τόσες ε, θέσεις οι οποίε δεν προσανατολίζονται στην ανάπτυξη. Οπότε ο προπολογισμό μα θα πρέπει να επικεντρώνεται ξεκάθαρα στην ανάπτυξη. Δηλαδή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, στην καινοτομία, στην έρευνα και να περιλαμβάνει λιγότερο άμεσες, λιγότερες άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο συνάδελφος από την Αυστρία μίλησε για ένα μέλλον στο οποίο θα έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών αυτός πρόκληση είναι ακόμα πιο μεγάλο από αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα έντονα, αλλά δηλαδή το θέμα της ε, απασχόλησης και της ανεργίας. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τα συνταξιδοτικά συστήματα, ώστε οι υγιείς ε, ηλικιωμένοι να έχουν κίνητρα για να συνεχίσουν την εργασία τους. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την, την ηλικία συνταξιοδότησης, να την επίπεδο στο ίδιο χρονικό ηλικιακό όριο με όλες αυτές τις εξελίξεις. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης ε, παράγοντες όπως οι γυναίκες ε, δεν εκμεταλλεύονται σωστά. Οπότε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την μελλοντική έλλειψη εργατικών χεριών θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην απασχόληση των γυναικών και θα πρέπει, όπως λέμε προηγουμένως, να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη γενικότερα. Όμως, αν θέλουμε να τα καταφέρουμε, τότε θα δούμε ότι τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι λιγότερο σημαντικά. Γιατί αρχικά θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ξαναλέω, στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που τρίσατε το χρόνο μιλή σα, λέει ο πρόεδρο. Ο, ο... Η ομιλία, συγγνώμη, ο λόγο τώρα. Ο λόγο στην κυρία Γιατούσκοβα από την ε, Τσεχία. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συγχαρώ την Βελγική Προεδρία και να την ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή συζήτηση αυτή για τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Γνωρίζω ότι και το Τσυχικό Κοινοβούλιο θα πρέπει αυτό να κάνει την ε, δουλειά του, να παίξει αυτό τον ρόλο του και πάρα πολλοί ε, ομιλητέ αναφέρθηκαν χθε στην ε, στρατηγική τη Λισαβόνα και ο κύριο Μπαρό αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και πάλι σήμερα το πρωί. Βεβαίω εμείς αποτύχαμε στο να πετύχουμε κάποιους από τους ε, στόχους ε, της Λισαβόνας. Όντως αυτό συνέβη. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας, αποφασίζοντας να εφαρμόσει την στρατηγική της Λισαβόνας έλαβε σημαντικές αποφάσεις. Μεταξύ άλλων να μην υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός σε θέματα που δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε. Η στρατηγική της Λισαβόνας μας έδειξε ότι η υπερβολική διάσταση και η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να είναι αναπόσπαστα στοιχεία της πολιτικής ανταγωνισμού μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να χτίσουμε τη στρατηγική μας πάνω σε αυτές τις βάσεις. Δεν θα πρέπει να έχουμε βεβαίως ανάπτυξη απλά και μόνο χάρη ανάπτυξεως. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να επικεντρωθεί σε αυτά τα δύο σημεία που σα ανέφερα. Και αυτό ακριβώς προσδοκά και ο υπόλοιπο κόσμο αλλά και οι πολίτε μας από εμά. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε. Η πολιτική της ε, Λισαβόνας, η πολιτική της Λισαβόνας, μάλλον η στρατηγική τη Λισαβόνας θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο επιτυχής εάν είχε εφαρμοστεί εξίσου ισχυρά σε εθνικό επίπεδο από ό,τι είχε εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Οπότε δεν θα πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος με τη στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να πετύχουμε ως μεμονωμένες χώρες αν κάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ε, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, όχι μόνο δίνοντας βεβαίως ας πούμε ε, κίνητρα φορολογικά, αλλά μέσω της βελτίωσης της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας κλπ. κλπ. Δηλαδή με άλλα λόγια με την προώθηση του κοινωνικού μοντέλου. Αυτά είχα να τονίσω και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που δώσατε την ευκαιρία στα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσουν με το Ευρωκοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρό της. Επειδή νομίζω ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, στην, ε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, το μέλλον της Ευρώπης θα εξαρτάται όχι πια από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μόνο, όσον αφορά την πρόθεση των κοινών μας στόχους, αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον επόμενο ομιλητή, στον κύριο Γιάν Κρέινερ από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες ιδέες όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Εμείς υπολογίζουμε νέους δείκτες και νέους τρόπους υπολογισμού αυτού του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ δηλαδή το απόλυτο χρέο σε σχέση με το ΑΕΠ στη χώρα μου είναι στο 70%. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο λογικό, γιατί το θέμα είναι γιατί δεν βάζουμε το δημόσιο χρέο σε μια θέση όπου θα συγκρίνεται με την ιδιωτική περιουσία στην κάθε χώρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό κατεβαίνει στο 22%. Ε, αν θέλετε λοιπόν να μειώσετε το δημόσιο χρέος στο 0, αυτό θα πρέπει να κάνετε. Αν δούμε λοιπόν τις, ε, τα περιουσιακά στοιχεία και την εξέλιξή τους ε, τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα μου, θα δούμε ότι είχαμε μια παρόμοια εξέλιξη ε, με αυτή που είχαμε σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και νομίζω σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν αρκετό να φορολογούσαμε κάτω από το 50% τη αύξηση τη ιδιωτική περιουσία και θα μειώνουμε κατά πολύ έτσι με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο χρέο. Οπότε νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αρκέσει. Θα αρκέσει να έχουμε ένα φόρο της τάξης του 50% όσον αφορά την αύξηση περιουσίας για να μην έχουμε καθόλου χρέο σε 10 χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερα χρήματα και με αυτόν τον τρόπο θα διοχετεύσουμε κεφάλαια και κονδύλια στην έρευνα και στην καινοτομία ώστε να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα ξεχνάμε όλα αυτά γιατί θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπία ε, στην κοινωνία μας μεταξύ παραγωγικότητας και δημοσίου χρέους επειδή οι κοινωνίες μας θα πρέπει, το ξαναλέω, να ε, εξορροπούν με αυτόν τον τρόπο που σας ανέφερα προηγουμένως την παραγωγικότητα και το δημόσιο χρέο. Ευχαριστώ να διαβάσω και λεπτομέρειε τι μου αυτέ στην Επιτροπή και όταν ακούμε από την Κομισιόν να γίνεται λόγο για αποπληρωμή δανείων κλπ. κλπ. Νομίζω θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα. Ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Αλμπέρτο Κώστα, από την Πορτογαλική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση νομίζω πρόσφατα ενσωμάτωσε την έννοια των συνετών πολιτικών. Δηλαδή μιας πολύ καλής ιδέας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς. Οπότε δηλαδή μπροστά σε προτάσεις ε, μεταρρυθμίσεων πολύ ενδιαφέρουσε και που υπόσχονται πολλά για το μέλλον όπως αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή εδώ βλέπουμε πολύ συχνά να υπάρχουν και μηνύματα λιγότερο συνετά να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο να πω το εξή για τις κυρώσεις. Μιλήσαμε για το κατά πώς θα πρέπει να υπάρχουν ή όχι κυρώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πολύ σημαντική και πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία. Θα ήταν όμως νομίζω συνετότερο εδώ να προβλέψουμε ένα σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Όμως δεν θα πρέπει τα, εθνικά κοινοβουλία απλά και μόνο να είναι θεατές των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πρώτο εξάμεινο. Δεν θα μιλήσω τώρα βεβαίω και για τα θέματα που αφορούν τη συνθήκη της Λισαβόνας και τα οικονομικά και την κατάσταση των οικονομικών. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε όργανα ή οργανισμούς που θα έχουν ουσιαστικό ρόλο, χωρίς δηλαδή νομοθετική αρμοδιότητα. Γιατί νομίζω ότι η νομοθετική αρμοδιότητα θα ακολουθήσει. Αλλά δεν θέλω να πει σε λεπτομέρειες. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το θέμα μιας ξαφνικής αναθεώρησης της συνθήκης μέσω δηλαδή απειλών για κυρώσεις ή ανατροπής Τη συνταγματική θέση μιας χώρα μέλου. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να υπάρξει συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι και τόσο συνετά ως αποφάσεις και προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς και τις ε, παράπλευρε απώλειε μετά από αυτέ τι μη συνετέ προτάσει και ιδέε που ακούσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφο. Επόμενος ομιλητής έχει το λόγο από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, κ. Καρίσου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο είναι τα θέματα που θέλω να θέσω. Το πρώτο είναι οικονομικού τύπου. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις οικονομίες των κρατών μελών. Το παράδοξο είναι ότι η κρίση αυτή και η έξοδος από την κρίση δεν θα λύσει το πρόβλημα αυτό της διαφοροποίησης και ίσως να μεγιστοποιήσει τις αποκλίσεις αυτές στον τομέα ιδιαίτερα της ανταγωνιστικότητας. Κάποιες χώρες, τόσο το καλύτερο για αυτές, έχουν περάσει σε διαδικασίες ανάκαμψης θεαματικής, άλλες είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα ανάκαμψης, χαρακτηρίζονται και από φαινόμενα ύφεσης. Ο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών λοιπόν, λοιπόν είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι επαρκή. Η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης θα πρέπει να αφορά και την μακροοικονομία και τα εμπορικά πλεονάσματα, έτσι ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει ένας πραγματικός συντονισμός. Αλλιώς οι διαφορές αυτές θα συνεχιστούν και στο τέλος θα απειλήσουν το ίδιο το ευρώ, το γνωρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έκανε μία πρόταση την οποία θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα, τη λεγόμενη μακροοικονομική εποπτεία. Στο τελευταίο συμβούλιο το θέμα αυτό, και ίσως να μην είμαι απόλυτα σωστά πληροφορημένος, δεν συζητήθηκε κατά προτεραιότητα και βασικό θέμα ήταν τα δημοσιονομικά. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής θα θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις αυτές με τη δημιουργία ενός πίνακα απόδοσης από ό,τι φαίνεται που ίσως θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και άλλα κριτήρια, να ανταλάβουμε υπόψη μας και όχι μόνο το κριτήριο του χρέους και το δημοσιονομικό και να υπάρξει μια μακροοικονομική συνεργασία ικανοποιητικότερη. Δεύτερη ερώτηση και τελειώνω. Ε, σχετικά με τη σύνδεση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, η πρωτοβουλία χθε και σήμερα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο επίσημη, πιο θεσμική. Έχουν γίνει ορισμένες προτάσεις για μια δημοσιονομική διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και αναρωτιέμαι πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας κάνει προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάρες. από την Άνω Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου Λόδος Χέσκινς. Θα ήθελα να μεταφέρω τις απόψεις μου στον τομέα του ενημέου νομίσματος πρώτα και στις κυρώσεις ε, κατά δεύτερον. Βασικό μάθημα της κρίσης είναι ότι απαιτείται για το ευρώ περαιτέρω πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω απόκλησης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης και για τις κυρώσεις. Η πιο ε, σοβαρή κύρωση για τις άτακτες χώρες είναι να ε, πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα ε, για να καλύπτουν τα έξοδα τους όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να δίδονται σωστές πληροφορίες στις οικονομικές αγορές έτσι ώστε να μπορούν να κρίνουν σωστά τις εθνικές οικονομίες πολύ νωρίτερα από τη στιγμή κατά την οποία το πρόβλημα θα είναι πλέον εκτός ελέγχου. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής από τη Φιλανδία, ένα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τον Βέλγο Πρωθυπουργό για τις εξαιρετικές τους παρεμβάσεις. Χαίρομαι διότι βλέπω ότι και το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή έχουν αναλάβει αυτή τη δέσμευση να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, χρειαζόμαστε κανόνες και για τις διεθνείς χρηματαγορές αλλά και για την, τις εσωτερικές στους, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να προβλέψουμε και να αποφύγουμε την επανάληψη της κρίσης του 2008. Θα πρέπει να ξανααποκτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στο ενιαίο νόμισμα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αρκετούς κανόνες μέχρι σήμερα. Το βασικό είναι να τους στηρίσουμε, να τους εφαρμόζουμε. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει πιο αποφασιστικά, να μεριμνήσει ώστε όλοι τηρούν τους κανόνες που έχουμε όλοι συμφωνήσει. Μόνο έτσι οικοδομείται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών αλλά και μεταξύ αγορών. Δεύτερο σχόλιο μου ε, είναι η ευθύνη των τραπεζών. Είναι σαφές ότι όντως ο χρηματοπιστωτικός κλάδος έχει πολλά κέρδη, συμμετέχει, ε, αναλαμβάνει κινδύνους. Και ίσως θα έλεγα ότι είναι αδύνατο ε, άλλες χώρες μόνο χωρίς τις τράπεζες να μπορέσουν να στηρίξουν τις υπόλοιπες χώρες ως προς τα ε, χρέη τους. Επομένως, στις μελλοντικές αποφάσεις σημασία θα έχει πιστεύω να τονιστεί η ευθύνη των τραπεζών. και των πιστωτών, εάν θα πρέπει να δοθούν νέες πιστώσεις τελικά για να στηριχθούν ορισμένα κράτη-μέλη. Το τρίτο σχόλιο μου έχει να κάνει με το φόρο στις ε, χρηματιστηριακές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές γενικότερα. Ε, όταν κανείς ταξιδεύει με αεροπλάνο ή με τρένο ή όταν κανείς μπαίνει σε ένα κατάστημα και αγοράζει κάτι, φορολογείται. Ο μόνος ε, χώρος, το μόνο πεδίο που είναι εκτός φορολόγησης είναι το πεδίο που έχει να κάνει με την κίνηση του χρήματος, την μετακίνηση των κεφαλαίων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε φόρο στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία από αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω διότι ούτε εσείς ε, ξεπεράσατε τα τρία λεπτά ακριβώς που είχατε στη διάθεσή σας. Γι' αυτό και περνούμε στον κύριο Edmund Βίτκουντ από την Πολωνική Γερουσία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πολλής λόγος έχει γίνει για τις απαραίτητες αλλαγές, για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, για να αποφύγουμε μία επανάληψη της κρίσης. Ας εξετάσουμε όμως το θέμα από διαφορετική σκοπιά και ας ε, τονίσουμε άλλους κινδύνους, άλλες απειλές. Ίσως ε, είναι σημαντικό να έχουμε νέα θεσμικά όργανα και νέες διαδικασίες εποπτείας. Αυτό λέμε. Κάποιοι όμως ειδικοί λένε ότι έχουμε αντιδράσει υπερβολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν φανεί κάποιες αδυναμίες ε, του συστήματος εποπτείας. Το εποπτικό σύστημα δεν λειτουργήσε ικανοποιητικά. Αυτό είναι σαφές. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν δώσουμε υπερβολικές αρμοδιότητες στις αρχές εποπτείας θα μπορέσουν ε, να ανταποκριθούν. Τελικά όλα αυτά τα συστήματα ε, διαχείρισης ε, έχουν ωφελήσει το καταναλωτή. Έρχονται σε αντίθεση με την ομοθεσία για τον ανταγωνισμό. η διαφορά μας ε, με την Ελβετία, αν θέλετε, ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει απαγόρευση αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, ε, σύμφωνα με ορισμένους οικονομικούς αναλυτές, οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται στο ρόλο αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν σε κάθε κράτος μέλος. Λόγω όλων αυτών των κινδύνων και των απειλών, Ορισμένα κράτη-μέλη αμφισβητούν αυτό το κριτήριο του 3% ε, και ζητούν ε, να ε, γίνει το ίδιο, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα που υπάρχει στι Πολιτείες όπου μπορούν, μπορεί να τυπωθεί χρήμα δισεκατομμύρια δολάρια για να διασωθούν συγκεκριμένες τράπεζες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Άλλωστε θα πρέπει να διδαχθούμε ε, από αυτά που γίνονται στη ΣΥΠΑ και ειδικά μετά, μετά τα αποτελέσματα στις ε, ε, ενδιάμεσες εκλογές στη ΣΥΠΑ στο μέσο της θητείας. Μήπως θα έχουμε τελικά υπερβολική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτός δηλαδή είναι ο κίνδυνος που θα ήθελα να σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάνν Μπόερ από την Τσεχία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Χαίρομαι που λαμβάνω εδώ το λόγο σήμερα. Ήμουν δήμαρχος παλαιότερα. Ξέρω ότι η εργασία που έχετε είναι δύσκολη και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μπαρόσο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Νομίζω ότι πολλές φορές οι φιλοδοξίε μας είναι τόσο μεγάλες που δεν επαρκεί ο προπολογισμό. Γι' αυτό ακριβώς τίνουμε να τον αυξάνουμε συνεχώς. Οπότε κύριε Μπαρόσο ρωτώ, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αυξήσουμε και πάλι τον ευρωπαϊκό προπολογισμό μέσω ιδιοπόρων ή μέσω νέων φόρων και ποιων φορών σε αυτή την περίπτωση. Επίσης να πω ότι στην Τσεχία και στο Τσεχικό Κοινοβούλιο είναι πολύ επίμαχο αυτό το θέμα των νεοφόρων. Δεύτερη ερώτηση. Στρατηγική. Από ό,τι ξέρω, η στρατηγική της Λισαβόνας δεν απετέλεσε μια επιτυχία. Μάλλον δεν ήμασταν σε θέση να ξεπεράσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής, οπότε η μου ερώτηση κύριε Μπαρόσο είναι το εξή. Η νέα στρατηγική 2020 θεωρείται, θεωρείται, λέω, ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε μεγαλύτερες ευθύνες οι οποίες θα απορρέουν από την επιτυχία ή αποτυχία της στρατηγικής αυτής 2020 να πω επίσης και κάτι άλλο. Δεν έχουμε τους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις ακόμα. Και στην περίπτωση της Ελλάδας ξέραμε ότι υπήρχαν προβλήματα εκ των προτέρων. Τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Όμως κανείς ειλικρινά δεν είχε την πρόθεση ή την όρεξη να εφαρμόσει κυρώσεις σε σχέση με τα χρηκονομικά κριτήρια. Ρωτώ λοιπόν για το μέλλον. Όταν θα έχουμε νέα χρηματοοικονομικά κριτήρια, όταν θα έχουμε κυρώσεις κλπ. κλπ. Τότε, κύριε Μπαρόζο, από ό,τι ξέρετε εσείς από τη δική σας εμπειρία, θα μπορούσαμε να βρούμε μια συνένεση συνένεση εδώ και να εφαρμόσουμε σωστά αυτές τις ε, κυρώσεις που τόσο συζητάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο πρώτο τελευταίος ομιλητής τώρα, ο Λόρδος Χάσκελ μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που διοργάνωσε αυτή την διάσκεψη. Συζητήσαμε πάρα πολύ το μέλλον και διαρωτώ με μήπως κατά λάθος ξεχάσαμε να εφαρμόσουμε κάποιους από τους υπάρχοντες κανονισμούς. Επί παραδείγματι, οι περισσότεροι από εμάς συμφωνούμε ότι ε, είναι θετική η νέα αγορά. Έχει πλεονεκτήματα για όλες τις χώρες μέλη. Και κάποιοι παραπονιούνται ότι κάποιοι από τους κανόνες, πολλοί κανόνες της νέας αγοράς δεν έχουν εφαρμοστεί. Εμείς λοιπόν ως Εθνικά, το Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν θα μπορούσε να μας ε, βοηθήσει εδώ πρακτικά ε, για να παροτρύνουμε τα συνδικάτα, τις επιχειρήσεις, όλους τους φορείς να διεκδικήσουν τα πλεονεκτήματα της ενίας αγοράς και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ώστε αυτά να εφαρμοστούν πλήρως. Επίσης νομίζω θα πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στους καταναλωτές όσον αφορά τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις δίνοντας έμφαση στις προεγραφές ποιότητας, μάλλον ασφάλειας στις ε, προδιαγραφές που αφορούν τις πρωτεσίλες ε, και να τονίσουμε γεγονό ότι αυτά τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας και αυτό ενδεχομένω να ήταν ένα πρακτικό μήνυμα το οποίο θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε στην χώρα μας και διερωτούμε κατά πόσο θα μπορούσε να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Ο λόγο τώρα στον τελευταίο ομιλώντα στον κύριο Μάσιμο και Καραβάλια από την Γερουσία την Ιταλική και να προχωρήσω και την προεδρία στον συνάδελφο Μαρτίνης Μαρτίνες. Έχετε το λόγο συνάδελφο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο θεματάκια. Πρώτη ερώτηση η Ιταλική Γερουσία υιοθέτησε ένα έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Μεταξύ των διαφόρων σημείων ένα σημαντικό από αυτά αφορά τους ε, πρόσθετους δείκτες που θα πρέπει να εξετάσουμε όταν αξιολογούμε τους προπολογισμού των διαφόρων χωρών μελών. Οι παραδοσιακοί δείκτες για τους προπολογισμού φαίνεται δεν λειτουργήσαν και επειδή είχαμε και τη σοβαρή οικονομική κρίση με αποτύπωμα στο χρέος, χρειάστηκε να κάνουμε αυτούς τους συμπληρωματικούς δείκτες. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε ας πούμε η συσσόρευση του ιδιωτικού χρέους, η καθαρή περιουσιακή θέση και επίσης η βιωσιμότητα κάποιων δαπανών όσον αφορά ας πούμε τις συντάξεις, παραδείγματος χάρη. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά αυτό που ήδη υπεθύμησαν οι Γάλλοι συνάδελφοι, δηλαδή την περασινή ιδέα του Λαμασούρ για μια επιτούτου διάσκεψη των ε, Επιτροπών Προπολισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επειδή όλες οι χώρες θα πρέπει να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις προτεραιότητες. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν και ακούστηκε αυτή η ιδέα για αυτή την διάσκεψη των Επιτροπών Προπολισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων που μας βρίσκει σύμφωνο και θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Επειδή θεωρούμε ότι μια τέτοια διάσκεψη υπομορφή απλή και άτυπη θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν και πιο λειτουργική από μια διάσκεψη τέλο πάντων πολύ επίσημη και διοργανωμένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, εκτενή κατάλογο, αλλά ευτυχώς όλοι τηρήσατε το χρόνο ομιλία σας. Οπότε, τώρα έχουμε τις δύο ομιλίες που θα σχολιάσουν τις ερωτήσεις. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπαρόσο για να σχολιάσει και να απαντήσει στα ερωτήματα που του απευθύνθηκαν ο προς της Κομισιόν. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πριν απαντήσω, μετά έτσι και θα έχει την ευκαιρία και ο κύριος Λετέρν να δώσει απαντήσεις, θέλω να τον συγχαρώ καταρχάς Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαι θα ευγνώμονες προς την Βελγική Προεδρία. Η Βελγική Προεδρία στα πλαίσια μιας ιδιαίτερα περίπλοκης κατάστασης την οποία βιώνουμε στην Ευρώπη σήμερα εργάζεται σκληρά, πιστικά και ήταν μεγάλη ευκαιρία για μας αυτή τη δύσκολη στιγμή της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, της θέσης ισχύ των νέων συνθήκων να έχουμε μια προεδρία τόσο ευρωπαϊκή, τόσο κοινοτική όσο η βελγική και τον Πρωθυπουργό Ιβ Λετέρνα. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν, πολλές από αυτές αφορούν τους φόρους, τα χρηματοπιστωτικά για την Λετωνή συνάδελφο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να υποστηρίξει πάντα την ιδέα ενός φόρου τέτοιου είδους συναλλαγών αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, σφαιρικά. Και εγώ αύριο θα πάω στη Σεούλ και αυτή θα είναι η θέση μου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας φόρος διεθνών συναλλαγών, διεθνής όμως, σφαιρικός. Εγώ νομίζω ότι να επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος μόνο στην Ευρώπη θα δημιουργηθούν προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Προσπαθούμε να δούμε άλλες δυνατότητες, τι έχουμε στη διάθεσή μας. Ο φίλος μας από τη Φιλανδία σαν παράδειγμα Νομίζω ότι παρουσίασε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βλέπουμε μερικές φορές ή να δημιουργείται η εντύπωση ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας μετέχει λιγότερο από άλλους τομείς στην προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη. Πέρα από το θέμα των τραπεζικών εγγυήσεων βέβαια, Υπήρξε ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρκετές επιλογές και ελπίζω να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις σύντομα σχετικά με τα, επιτόκια, με τα ποσοστά επιβολής φόρου. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητήσουμε και ελπίζω να εγκρίνουμε ένα πακέτο για ε, υποδομές στον τομέα της ενέργειας και θα επισημοποιηθεί η απόφαση την επόμενη Πέμπτη. Είναι μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της ενέργειας και τι κοινή πολιτική μπορούμε να ακολουθήσουμε. Για τον Πολωνό συνάδελφο υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από την Πολωνία. Αυτό δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον και αφοσίσωση της Πολωνίας στην προσπάθεια που κάνουμε για τον σωστό συντονισμό των νομικών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να έχουμε μια πλήρη εναρμόνιση στην Ευρώπη του φορολογικού συστήματος. Εγώ δεν σας λέω κάτι. Το μυστικό στο τελευταίο Συμβούλιο ένα κράτος μέλος πρότεινε μια συγκεκριμένη διατύπωση σε σχέση με ένα κοινό φορολογικό ποσοστό κτλ και υπήρξε μια απόρριψη θα έλεγα πολύ ε, ξεκάθαρη από τις περισσότερες άλλες χώρες. Αυτό που είναι χρήσιμο όμως για τις επιχειρήσεις μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα είναι να υπάρξει μια κοινή φορολογική βάση και σωστή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μια κοινή επιχειρηματική φορολογική βάση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ευκολότερες για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάποιοι από αυτούς που έθεσαν ερωτήσεις δεν είναι παρόντες, αλλά θα ήθελα να δώσω κάποιες συνοπτικές απαντήσεις. Στο Λόρδο Χάσκελ, σαν παράδειγμα, να πω ότι μία από τις βασικές μας ανησυχίες μας είναι το πώς μπορούμε να πείσουμε το ευρωπαϊκό κοινό. Και γι' αυτό και ζήτησα από τον μόνι να μας προετοιμάσει μια έκθεση για την εσωτερική αγορά. Συμφώνησε. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες της Ένωσης ε, δεν ερωτεύονται την εσωτερική αγορά, ίσως σε κάποιες χώρες. Πρέπει λοιπόν να συμφιλιώσουμε την ιδέα της αγοράς με τον πολίτη μέσω της κατανάλωσης, μέσω της ιδιότητας του καταναλωτή που έχει ο πολίτης. Η λογική της ενιαίας πράξης για την εσωτερική αγορά είναι να μην υπάρχουν εμπόδια, να ολοκληρωθεί φυσικά η εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα να υπάρξει πολιτική στήριξη από πλευρά των εμπλεκομένων γι' αυτό. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε μια τέτοια αγορά πλήρη στην Ευρώπη. Σε κάποιους τομείς έχουμε, αλλά όχι συνολικά και δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι προς τα έξω όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες που απαιτούνται στο εσωτερικό μας. Πώς μπορούμε να συνομιλούμε σαν παράδειγμα με κάποιους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό και να τους ζητάμε ότι θα πρέπει να σέβονται την εσωτερική μας αγορά όταν εμείς ακόμα δεν την έχουμε ολοκληρώσει. Το θέμα λοιπόν είναι σημαντικό για μας και θα επιμείνω σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Λόρδος Χάσκελ. Το θέμα είναι να εφαρμόσουμε σε μια πρώτη φάση ε, τις αποφάσεις και τα πλαίσια που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό εμείς ξεκινάμε διαδικασίες επί παραβάση και παραλήψη εναντίον όλων των χώρων που δεν σέβονται τις βασικές αρχές της εσωτερικής αγοράς. Έχω μια εμπειρία 6 ετών τώρα. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα υπήρχε ουσιαστικά εσωτερική αγορά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ενιαία αγορά. γιατί συνεχώς θα ζητούνται εξαιρέσεις, παρενθέσεις, προσωρινές απαλλαγές και αυτό θα λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος και στο Ηνωμένο Βασιλείο να κατανοήσει ο κόσμος ότι για να υπάρξει μια τέτοια αγορά απαιτεί θεσμικά όργανα. Η δημιουργία μιας αγοράς είναι μια θεσμική δημιουργία ουσιαστικά και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα είναι σημαντικός αν θέλουμε να υπάρξει ενιαία αγορά, να αναπτυχθεί ενιαία αγορά, να ευαθυνθεί ενιαία αγορά και οι προτάσεις που κάνει ο Λόρδος Χάσκελ είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές. Αυτό κάνουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε και σε εθνικό επίπεδο να δείξουμε τι είναι η εσωτερική αγορά, τι προσφέρει στους Ευρωπαίους η εσωτερική αγορά, γιατί πολλές φορές νέοι ιδιαίτερα Το μόνο που θέτουν ε, θα έλεγα είναι το θέμα της δίκαιης επιστροφής. Πόσα δίνω, πόσα παίρνω. Όσοι περιορίζονται σε τέτοιου είδους λογαριασμούς είναι αυτοί που ωφελούνται από την εσωτερική αγορά, αλλά το ξέρουν αυτό. Ξέρουν πόσο τους βοηθάει ας πούμε στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης η εσωτερική αγορά. Και η συζήτηση η οποία θα γίνει για τις δημοσιονομικές προοπτικές νομίζω θα δείξει ακριβώς ποια είναι η αξία της εσωτερικής αγοράς. Η ερώτηση του εκπροσώπου της Τσεχικής Βουλής Μπάουερ αν καλά. Συνειδητοποιούμε την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη σήμερα και ακριβώς λόγω ακριβώς των συγκεκριμένων περιορισμών των δημοσιονομικών των εθνικών έχουμε θέσει το θέμα προσυζήτηση το θέμα προσυζήτηση των ιδίων πόρων. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες δαπάνες. Ακριβώς επί τα κράτη-μέλη έχουν δυσκολίες να κρατήσουν το ίδιο επίπεδο συνεισφοράς προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στον τομέα των ιδίων πόρων όπως το προέβλεπε η συνθήκη της Ρώμης, λέει ο μιλητής. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η στιγμή. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για φόρους, είναι δύσκολο να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Αν θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους, χρειάζονται μέσα και οικονομικά μέσα. Ελπίζω λοιπόν με επικοδημητικό τρόπο να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ελπίζω να αποκλείσουμε τάσεις εθνικιστικές και λαϊκιστικές από τη συζήτηση αυτή. Αν ο ευρωπαϊκό προπολογισμό αντικατοπτρίζει μόνο αυτά τα οποία λέγουν οι εθνικοί προπολογισμοί, αυτό δεν είναι αληθέ. Ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι εντελώ διαφορετικό από του εθνικού προπολογισμού. Καταρχά δεν υπάρχει χρέο, α πούμε, στο επίπεδο ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει χρέο. Και οι εθνικοί προϋπολογισμοί εδώ πρέπει να κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια γιατί πολλές χώρες ε, συνεχίζουν να λειτουργούν με πάρα πολύ ε, υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μπορεί να ισχύει, αλλά ισχύει για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στον ευρωπαϊκό δεν ισχύει. Ε, μια άλλη διαφορά είναι ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, σαν παράδειγμα, οι πιο πολλοί, οι δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% ή και πάνω από 50% οι τρέχουσες δαπάνες του ΑΕΠ για τη λειτουργία του κράτους, για την κοινωνική πρόνοια κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αντίστοιχο προϋπολογισμό μιλάμε για 5,7, 5,8%. Το διοικητικό κόστος δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα τα υπόλοιπα στον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι επενδύσεις επενδύσεις στις πολιτικές, στη γεωργία σαν παράδειγμα, στη συνοχή και σε νέους συνεχώς τομείς. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δημιουργήσει νέες δομές, νέες δραστηριότητες όπως την εξωτερική υπηρεσία δράσης. Πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, οι στιγμές είναι δύσκολες και μερικές φορές όταν υπάρχουν κάποια επιχειρήματα εθνικά δεν αφήνουν χώρο να ακουστούν άλλα επιχειρήματα. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να φανούμε λογικοί, κατανοούμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά και πολιτικά σε διάφορες χώρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να σταθούμε κοντά ο ένας τον άλλον και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Σε ορισμένους τομείς η ευρωπαϊκή διάσταση προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ό,τι οι εθνικές προσπάθειες. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινεί. Την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όταν τα συζητάμε όλα αυτά με τους Αμερικανούς φίλους, τους Ρώσους, τους Κινέζους κτλ, όπως θα γίνει τώρα στη συνάντηση της ομάδας των 20, αν δεν συνεργαστούμε η δυνατότητα μόχλευσης των πραγμάτων που θα έχουμε θα είναι ελάχιστη και σε οικονομικό και σε δημογραφικό και σε πολιτικό επίπεδο η επιρροή μας θα είναι μικρή. Δεν θα επηρεάσουμε ουσιαστικά την παγκόσμια συζήτηση. Σήμερα όμως μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να προκαλέσουμε αλλαγές στην κατάσταση εφόσον θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες και στα πλαίσια της σωστής εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς και στα πλαίσια της μη αμφισβήτησης της εσωτερικής αγοράς και στα πλαίσια της εκμετάλλευσης όλων των πολιτικών συντονισμού που έχουν γίνει τώρα. Στην ερώτηση του Λόρδου Χάσκινς. Ενίο νόμισμα σημαίνει περισσότερη οικονομική διακυβέρνηση. Προφανώς. Και γι' αυτό είδαμε που είχαμε δυσκολίες και ακριβώς ενισχύουμε τη λεγόμενη οικονομική διακυβέρνηση. Έχουν υπάρξει ιδέες πολλές, το ευρωπαϊκό εξάμεινο κτλ. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια ουσιαστική συντονιστική δράση στον τομέα της οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει. Τι συνέπειες θα υπάρχουν για τα κράτη-μέλη εξ αυτού. Καταρχά, οι περισσότερε από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να μπουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μόνο οπτά ότι υπάρχει, μια εξαίρεση. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά όλε οι άλλε χώρε στην ουσία προσαρμόζουν τι πολιτικέ του με τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Μεγάλη Βρετανία, και δεν είναι μέλο της ζώνης, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει κάθε συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Είτε μας αρέσει είτε όχι λοιπόν. Είμαστε πολύ περισσότερο εξαρτημένοι σήμερα από ό,τι στο παρελθόν, με ή χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τα χρέη τα οποία έχουν Άλλες χώρες δεν έχουν ε, τα προβλήματα αυτά ή αν τα έχουν δεν είναι στη ζώνη ευρώ. Συνεπώς λοιπόν η κατάσταση δεν εξηγείται από το να είναι κανείς στη ζώνη ή να μην είναι στη ζώνη ευρώ. Το θέμα είναι η σημερινή μορφή της διεθνούς οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας και οι πολιτικές οι οικονομικές οι οποίες ακολουθούνται, οι δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται, οι οποίες σε πάρα πολλές από τις χώρες μας ήταν πράγματι μη υποστηρίξιμες. Πολλοί διαμαρτύρονται για τις αγορές, για την κατάσταση που υπάρχει κτλ. Προφανώ, όποιο δεν έχει χρέο δεν πηγαίνει, δεν προσφεύγει στι αγορέ, στι χρηματαγορέ. Το θέμα είναι να δούμε όμω τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικονομικών μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε να καταστήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστική. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε και στο θέμα των κυρώσεων. Λόρδος Χάσκινς επίσης και σωστή και διαφανής ενημέρωση. Προφανώς αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Στα πλαίσια της προηγούμενης Επιτροπής είχαμε ζητήσει περισσότερες αρμοδιότητες για τη Eurostat, για την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, για να ελέγχει τα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Απερίφθη η πρόταση αυτή γιατί είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα παρεμβατική. Η πραγματικότητα για την ελληνική περίπτωση ήταν ότι τα δεδομένα που παίρναμε από την Ελλάδα δεν ήταν τα κατάλληλα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Τώρα όμως έγιναν νέες προτάσεις, έγιναν νέες προτάσεις και τι εγκρίνουν τα κράτη-μέλη χωρίς διαφάνεια στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, το σύστημα δεν θα δουλέψει. Ούτε η νομισματική ένωση, είτε οποιαδήποτε άλλη αγορά. Απαιτούνται διαφανείς διαδικασίες ενημέρωσης ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το πετύχουμε αυτό. Είναι προς το συμφέρον όλων. Για τον συμπατριώτη μου, τον κύριο Κώστα. Πράγματι, ε, σχετικά με το πόσο επιφυλακτικοί και προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα έχει φανεί ιδιαίτερα επιφυλακτική, ιδιαίτερα όταν κάνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στη συνθήκη, αναθεωρήσεις της συνθήκης. Εδώ ίσως ο συνάδελφος Λετέρμε μπορεί να σας δώσει καλύτερες ε, εξηγήσει για το ποιε είναι οι θέσει των κρατών μελών. Το θέμα είναι ότι πράγματι συμφώνησαν τα κράτη-μέλη ότι υπάρχει ανάγκη ενό μόνιμου μηχανισμού απάντηση στην κρίση. Και χωρί τη Γερμανία αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Στη γερμανική περίπτωση πράγματι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια μεταρρύθμιση της συνθήκης για να διαρρυθμιστεί ένα θέμα το οποίο θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό για τη Γερμανία ακόμα και σε νομικό επίπεδο οι νομομαθείς φίλοι θεωρούν ότι η θέση αυτή των Γερμανών δεν είναι ένα καπρίτσιο δικό τους, είναι μια πραγματική ανάγκη. Και γι' αυτό ακριβώς μετά από τις γερμανικές προτάσεις τα κράτη-μέλη συμφώνησαν. Κανένας βέβαια δεν τρελαίνεται από την ιδέα να αλλάξει συνθήκη. Κανένας δεν ήταν ενθουσιώδης με την γερμανική πρόταση, αλλά παρόλα αυτά δεχόμαστε τη λογική να υπάρξει μια περιορισμένη αναθεώρηση της συνθήκης πλέον. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι όλα τα κοινοβούλια θα πρέπει να εκ να εκφραστούν γιατί πρέπει να υπάρξει επικύρωση από τα 27 κράτη. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη και για τα κοινοβούλια να εκφραστούν για μια ακόμη φορά. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας κύριε Κώστα. Υπάρχει η πρόταση να χρησιμοποιήσουμε το νέο σύστημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Αυτό μπορεί να γίνει και μαζί με την ΚΟΣΑΚ. Η συναδρίαση της ΚΟΣΑΚ τον Μάιο που θα γίνει στην Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτού του εξαμήνου ή της ετήσιας βάσης κοινοβουλευτικής συνεργασίας θα δούμε. Έτσι ώστε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε καλύτερα τα κοινοβούλια των κρατών μελών σε αυτή την προσπάθεια. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θα ήθελα να πω ποια είναι η άποψή μου. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας είχαμε ξεκινήσει μια ανεπίσημη συνεργασία με ανταλλαγή απόψεων κτλ. Παρ' όλα αυτά ένα πράγμα θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα βαρύ και πολλές φορές ιδιαίτερα αργό. Πρέπει εμεί να εφαρμόσουμε βέβαια αυτά τα οποία υπάρχουν στη συνθήκη. Δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε νέε δομέ για τη λήψη επίσημων αποφάσεων. Υπάρχει ο μηχανισμό. Η Επιτροπή προτείνει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που συναποφασίζουν στι περισσότερε περιπτώσει. Εσεί τα εθνικά κοινοβούλια ελέγχετε τι δικέ σα κυβερνήσει. Αυτή είναι η βασική σα αρμοδιότητα. Πέραν αυτού τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει ορισμένες νέες διαδικασίες, όπως το θέμα του ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας. Αυτό το οποίο βλέπω εδώ και απαντώ ήδη και στις ερωτήσεις άλλων συναδέλφων του κυρίου Καρέσα από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Υπάρχει δυνατότητα με ανεπίσημο τρόπο να ξεκινήσουμε μια μορφή στενή συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράδειγμα, δημοσίευσε πρόσφατα, στις 27 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα εργασίας της για το 2011. Παρουσιάζει ένα πλήρη κατάλογο όλων των σχεδίων τα οποία θα προωθήσουμε το 2011, ακόμα και για το 2012. Ε, είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια εφόσον το επιθυμούν να ξεκινήσουν να συζητούν άμεσα τους τομείς τους οποίους σκοπεύουμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρξει εμπλοκή σας, πρέπει να νιώσετε κι εσείς ότι σας αφορά αυτή η διαδικασία. Ας μην είμαστε τόσο θεσμικοί πέραν αυτών των θεσμών που ήδη λειτουργούν μέσω της συνθήκης. Και μιας και αναφερόμουν σε αυτά που έλεγε ο κύριος Καρές να συμπληρώσω λέγοντας ότι οι προτάσεις που έχουν γίνει σχετικά με τη μακροοικονομική επίβλεψη και τις προτάσεις για τη μακροοικονομική επίβλεψη είναι τμήμα των προτάσεων τις οποίες έχει ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και μετά από τις προτάσεις και της Επιτροπής Βαν Ρόμπαϊ έχουν υπάρξει ε, συζητήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν θέλει θα υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές. Αλλά είναι στο κανονικό θα έλεγα δίκτυο, θα έλεγα το νομοθετικό. Λοιπόν, ναι, συντονισμός στις οικονομικές πολιτικές. Εδώ υπάρχει από τη μία η οικονομική και νομισματική ένωση, αλλά ε, δεν είναι μόνο νομισματική ένωση είναι οικονομική και νομισματική και σημασία έχει περισσότερο το οικονομικό παρά το νομισματικό. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι επαναστατικό, με την καλή έννοια επαναστατικό. Θα υπάρξει ένα σύστημα πολύ πιο ολοκληρωμένο. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταργηθούν θα πρέπει να απορριφθούν από μια ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προχωρήσει πολύ σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σε σχέση με τον καλύτερο συντονισμό. Και το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα έλεγα είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο σέβεται τις αρμοδιότητες των, των εθνικών κοινοβουλίων. Οι προτάσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές επί τη βάση της εκθέσεως Λαγοζιέ και έχουν γίνει δεκτές και από το Κοινοβούλιο και ομόφωνα από το Συμβούλιο να υπάρξει ένα σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρώπη. Πριν δύο χρόνια άμα έλεγε κανείς κάτι τέτοιο δεν θα το θεωρούσε κανείς δυνατό. Σοβαρά. Βλέπετε λοιπόν ότι καθημερινά τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η τάση και να δούμε ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία απαιτεί η κρίση με τα μέσα τα οποία έχει. Μερικές φορές είναι κοινοτικά τα μέσα αυτά, μερικές φορές είναι διακυβερνητικά τα μέσα αυτά, αλλά παρόλα αυτά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίνει να γίνεται συστηματικά πιο συνεκτική και διαρθρωμένη. Μίλησα πάρα πολύ ώρα, αλλά μου θέσατε και πάρα πολλές ερωτήσεις. <coughs> Μία τελευταία ερώτηση σχετικά με τη στρατηγική 2020. Ερώτηση από τον Τσέχο φίλο. Η πραγματικότητα της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν ότι ήταν καλή στρατηγική. Αλλά υπήρχαν προβλήματα εφαρμογής, ιδιαίτερα εμπλοκής σε εθνικό επίπεδο. Με το νέο σύστημα διακυβέρνησης αν οι κυβερνήσεις σας, αν τα κοινοβούλια σας συνεργαστούν, τότε θα πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η ειλικρινή μου άποψη, έχοντας βιώσει τα τελευταία έξι χρόνια σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παλαιότερα σαν Πρωθυπουργό στη χώρα μου. Μπορούμε να καταστήσουμε επιτυχή την ατζέντα τη Λισαβόνας, εξαρτάται όμως από τη δική σας προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους όλοι έχουμε θέσει για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς πολύ καλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως μιλήσατε πολύ, αλλά μιλήσατε και πολύ καλά. Και νομίζω ότι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 να εκφράσω την απόλυτη συμφωνία μου και τη στήριξή μου ε, στα λεγόμενα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετικά δραστήρια, εξαιρετικά ενεργητική και είναι έτοιμη να απαντήσει, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό το ότι εμείς ως Ευρώπη είμαστε παρόντες και προσφέρουμε απαντήσεις στη μεγαλύτερη κρίση που έχει σημειωθεί ε, αυτή των τελευταίων χρόνων μεγαλύτερη από το, ε, από το 1929. Ας μιλήσουμε τώρα για τον φόρο των χρηματιστηριακών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Ε, υπάρχει φάκελος ε, για το θέμα αυτό και σε επόμενο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ κρατών μελών. Τώρα, ως προς τον προϋπολογισμό, θα πρέπει τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και που έχουν και οι κρατικές αρχές και οι υπηρεσίες στη διάθεσή τους να τα ε, αξιοποιήσουμε στο μέγιστο για την οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε το όργανο της ευελιξίας 0,03% αν δεν απατώμε του ΑΕΠ που μπορεί να δοθεί ε, ε, σε προτεραιότητες οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με την αναγκαιότητα της στιγμής. Υπάρχει δηλαδή αυτό το εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό και η Βελγική Προεδρία αυτή τη στιγμή καταρτίζει προτάσεις ε, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη οι οποίες ή θα εγκριθούν ομοφόνος ή θα εγκριθούν με τη διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας για να αξιοποιηθεί ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο αυτό το εργαλείο ευελιξίας που έχουμε που μας επιτρέπει να αξιοποιούμε κονδύλια ε, προς όφελος της πολιτικής για την ανάπτυξη. Τώρα, ως προς την οικονομική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία που έχει αυτή η στρατηγική. Πριν από 1,5 μήνα νομίζω ότι ε, συζητήσαμε εκπάθρον το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Πρωθυπουργό χώρας μέλους και ως Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή έχω να σας πω ότι είναι ζωτική σημασία η στρατηγική αυτή να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να εφαρμοστεί πάνω σε στέρεα θεμέλια. Και γι' αυτό Έχουμε δουλέψει πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε συμφωνήσει ότι τα χρονοδιαγράμματα θα είναι εξαιρετικά αυστηρά και θα τηρηθούν απαρεγκλήτως. Και είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνουμε και με τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή, η πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 πρέπει να έχει κοινωνική διάσταση βάσει των στόχων που έχουν τεθεί από εσάς και θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να τονίσουν τη σημασία που έχει μια τολμηρή ε, πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα βιομηχανική. Δηλαδή, σε αντίθεση ε, με τον αγγλοσαξονικό κόσμο ή τον αμερικανικό κόσμο, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε και το βιομηχανικό βραχίωνα ε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τολμηρή ε, βιομηχανική πολιτική και αυτή η πολιτική μπορεί να ε, παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο και πρωταγωνιστικό ε, όταν γίνεται λόγος και για τις βασικές πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες φάρους. Τώρα, ως προς την εποπτεία, τον, τη χρηματοπιστωτική εποπτεία θα, καλό θα είναι να διδαχθούμε όλοι από τα μαθήματα που υπάρχουν στα συμπεράσματα της ειδική ομάδας που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ώστε να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατό τα επιπρόσθετα αυτά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μετά από τα συμπεράσματα, αυτά τα συμπεράσματα ουσιαστικά θα μεταφραστούν σε νομοθετική πρωτοβουλία ε, την οποία και θα εξετάσουμε και θα υιοθετήσουμε στη συνέχεια για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, ε, ε, αρνητικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη σημασία της πράξης για την ενιαία αγορά όντως υπάρχουν κάποια εμπόδια στην λειτουργία της ενιαίας της εσωτερικής αγοράς, υπάρχουν κάποια τέλματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και έχουμε αναγνωρίσει, άρα θα πρέπει να πείσουμε και την κοινή γνώμη η οποία συχνά δεν συνειδητοποιεί τι σημαίνει αυτή η αίσθηση του ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, ο κόσμος κάνει ουρά ε, για να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρίτες χώρες και εμείς που είμαστε μέσα, οι πολίτες μας που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά ε, δεν συνειδητοποιούν πόσα ωφέλη έχουν ε, στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο διότι είναι πολύ χρηστικό το ενίο νόμισμα, αλλά διότι αποκτούν προστιθέμενη αξία με αυτό το κοινό οικονομικό εγχείρημα. Και εμείς λοιπόν ως πολιτικοί ηθήνοντες θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να πείσουμε περισσότερο ε, την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για τα ωφέλη του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξέρετε, στην οικονομία ένα και ένα δεν κάνει δύο, κάνει παραπάνω από δύο. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε οικονομικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχουν πολλαπλασιαστικά ε, θετικό αποτέλεσμα. Για να ολοκληρώσω κάπου εδώ θα έλεγα ότι το οικονομικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται καταρχάς στην πρόληψη ούτως ώστε να μην επαναληφθεί τέτοιου είδου ε, κρίση, κατά δεύτερο λόγο στην ενίσχυση των οικονομιών. Όλα αυτά τα έχουμε δρομολογήσει και θα ήθελα να πω ότι τόσο οι κυβερνήσεις όσο τα κράτη-μέλη, όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ο πολίτης όλοι βασιζόμαστε σε αυτή τη συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε γρήγορα να εφαρμόζονται οι αποφάσεις που έχουν υιοθετηθεί ε, βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχα να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων η οποία ήταν πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λετέρν, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Βελγική Προεδρία και να παραλάβω τις λέξεις του Προέδρου, τα λόγια του, για το κατά πόσο δηλαδή είναι αξιοθαύμαστη και αξιοσημείωτη η προσπάθειά σας. Βλέπουν και οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια μέχρι ποιου σημείου ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις τα ευρωπαϊκά μεταξύ τους, όταν βέβαια αυτό είναι δικαιολογημένο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από αυτές τις δύο θαυμάσιες ομιλίες του Προέδρου της Κομισιόν και του Προέδρου του Συμβουλίου, θα μπούμε στην τελευταία φάση, στην φάση των συμπερασμάτων, με μια ομιλία του Συμπροέδρου μας, του κ. Ντεμεγέρ, και μετά θα έχουμε τα τελευταία λόγια ο πρόεδρο τη Βελική Γερουσία, κ. Ντεμέγερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καταρχήν δύο λόγια για να σας πω ότι ως αντιπρόεδρος του Βελγικού της Βελγικής αλλά και ως ε, δήμαρχος έχω πολύ φιλοευρωπαϊκά αισθήματα και με τιμά η παρουσία σήμερα εδώ και θεωρώ ότι πραγματικά βρισκόμαστε στο σπίτι της Δημοκρατίας Ευρώπης. Συμμετείχαμε σε μια ανοιχτή συζήτηση, πλούσια, ακούσαμε ε, τρεις υψηλού επίπεδου εισηγητέ σε σχέση με τις ε, εργασίες που έγιναν στις ομάδες χθες. Ο Μπρονο Τόιμπενς, συνάδελφος και συμπατριώτης, μίλησε για την κατάσταση απασχόλησης στην Ευρώπη το αύριο. Η Ευρώπη και το μέλλον της οικονομίας βρίσκεται στην ε, πράσινη οικονομία και στην ε, έρευνα μα είπε η κρίση δεν πέρασε ακόμα αλλά θα πρέπει βέβαια να ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε μάλλον την εξέταση του μέλλοντο, το πώ θα έχει το μέλλον δηλαδή για την στρατηγική μας. Η κυρία Μπερέ μίλησε για εκ μέρου της ομάδας εργασία που ασχολήθηκε με τη μελλοντική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και μας είπε ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το πιο σημαντικό επίπεδο διακέβρινσης. Μας είπε όμως και για την συμμετοχή των, Εθνικών Κοινοβουλίων και των Ευρωπαϊκών Οργάνων ώστε να τονώσουμε τις ε, και να ανταποκριθούμε στις εθνικές ευαισθησίες και αυτό θα είναι πάρα πολύ εύκολο έργο. Ο κύριος ε, Βιλαζόνα ο συζητητής της τρίτης ομάδας εργασίας τόνισε τη σημασία ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, της ενίσχυσής της και της προώθησής της στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Ένωσης. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι σημαντική στο πλαίσιο αυτό, λόγω της σημασίας του τομέα των υπηρεσιών στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Οπότε η γραφειοκρατία θα πρέπει να αποφευχθεί, μας είπε, και ούτως ή άλλως, αν αυτό δεν γίνεται, να μειωθεί σημαντικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω ότι με μεγάλη χαρά άκουσα τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος με τον ενθουσιασμό που τον διακρίνει υπενθύμησε τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της κρίσης. Δεν βρισκόμαστε στο τέλος της, αλλά με τον μεγάλο έλεγχο των αγορών, οικονομικών αγορών και με τα φιλόδοξα σχέδια Τη Στρατική 2020 μας είπε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Να πω εδώ ότι έχω την αίσθηση ότι η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Πρόεδρό της θα είναι θετική για να αναζητήσουμε λύσεις βιώσιμες και συνεπείς στην οικονομική κρίση. Και θα πρέπει να σας πω ότι άκουσα τις απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν και αυτό το κάνουμε μεγάλη χαρά. Ο κύριος Λετέρν, ο πρωθυπουργό μου, ως προεδρεύων, γνωρίζει πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωρίζει την ανάγκη καταπολέμησης της κρίσης μέσω ελέγχου των χρηματοπιστωτικών αγορών της στρατηγικής 2020, της ε, Ευρώπης ε, της αριστείας κλπ. κλπ. Τα λόγια του είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν πραγματικότητα χάρη στις κοινέ μας προσπάθειες. Η συμφωνία που είχαμε πρόσφατα καταδεικνύει ότι με την Νότιο Κορέα καταδεικνύει ότι η συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες αλλά και με τις μακρινές χώρες θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην επίλυση της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Τέλος, θα έλεγα ότι η σημερινή μας συζήτηση καταδεικνύει το γεγονός ότι όλοι μας, βουλευτές, κυβερνήσεις, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είμαστε έτοιμοι με πεποίθηση και επιμονή να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση και με χαρά βλέπω ότι πέραν των προσωπικών μας ευαισθησιών υπάρχει συνένεση για το, για το κύριο μέρος των πολιτικών που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτά, Πρόεδρε, εγώ είχα να πω ως συμπεράσματα μετά από αυτές τις συνεδριάσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Οι ομιλίες του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, του Πρόεδρου της Κομισιόν και ιδιαίτερα η ομιλία του συναδέλφου, φίλου και συντρόφου κ. Ντεμεγέρ επιτρέπει σε μένα προσωπικά να ολοκληρώσω την συνεδρίαση αυτή και να μην αφιερώσω καθόλου χρόνο στην ανάλυση των συμπερασμάτων και στο περιεχόμενο των συζητήσεων που έγιναν. Οι εισηγήσεις από τις ομάδες εργασίας έχουν ήδη διανεμηθεί, νομίζω οι δύο από τις τρεις. Η τρίτη ε, συντάσσεται και θα σας διανεμηθεί σε όλους. Εγώ θα αφιερώσω τα 4-5 λεπτά που θα χαρίσω στον εαυτό μου στα πλαίσια της διαδικασίας για να σχολιάσω κάτι το οποίο θεωρώ κεφαλαίου σημασία και που ανακύπτει από αυτή την συνεδρίαση. Καταρχήν θα ήθελα η Γκάρδια να χαιρετήσω τον ευχάριστο επικοδομητικό τρόπο γεμάτο έμπνευση που διέπει τις συνεργασίες και την επαφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια, με τις Γερουσίες, Βελγικό Κοινοβούλιο και Γερουσία κτλ. Ακούσαμε τα συγχαρητήρια προς την Κομισιόν για την διεργάνωση της συνάντησης αυτής. Όμως να σας πω ότι η συνάντηση αυτή διεργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα δύο σώματα του Βελγίου. Θα πρέπει λοιπόν να συγχαρούμε αυτούς ακριβώς τους παράγοντες και τους υπαλλήλους βεβαίω τους υπαλλήλου των δύο βουλών του Κοινοβουλίου και τους υπαλλήλου του Ευρωκοινοβουλίου, οι οποίοι τέλος πάντων συνέβαλαν επιμελητιακά και μας επέτρεψαν να εργαστούμε με τρόπο ικανοποιητικό που νομίζω ότι τελικά εργαστήκαμε. Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω το εξή σχόλιο. Τη σημασία δηλαδή που έχει αυτή τη στιγμή η απαραίτητη συνεργασία Ευρωβουλής Εθνικών Κοινοβουλίων, κάτι το οποίο ήταν πάντοτε επιθυμητό. Μετά όμως την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, της νέας δηλαδή πολιτικής και νομικής βάσης, επί της οποίας θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχασε 10-15 χρόνια αμφαλοσκόπησης και αφού παρέλειψε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μας κάνει ένα παγκόσμιο παίχτη και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από την οικονομική υπερίσχυση και όχι από τις πολιτικές τάσεις. Σε αυτή λοιπόν τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνεται η υποχρέωση συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια και περιλαμβάνεται επίσης κάνοντας μία συγκεκριμένη στα εθνικά κοινοβούλια γύρω στις 14 φορές στη συνθήκη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτή η εμπειρία που συλλέγουμε και εγώ ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου έχω το χαρτοφυλάκιο των σχέσεων ευρωβουλης Εθνικών Κοινοβουλίων και υπάρχουν και άλλοι δύο συνάδελφοι οι οποίοι με στηρίζουν σε αυτήν την εργασία. Να πω λοιπόν ότι εμείς είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία οι 27 χώρες μέλη για το κείμενο της Εθήκης Λισαβόνας. Από τη στιγμή όμως που υπήρξε πολιτική συμφωνία ήταν σχετικά εύκολο να συνταχθούν διάφορα άρθρα και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιο περίπλοκο να μεταφερθούν στην πράξη και να εφαρμοστούν δηλαδή αυτές οι παράγραφοι των άρθρων της συνθήκης. Και εδώ ακριβώς αντιμετωπίζουμε σχετικά δηλαδή με την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων σε όλη την διαδικασία των, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από την εκπόνηση και σύνταξη μέχρι την εφαρμογή. Εκεί λοιπόν βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που βεβαίως προσπαθούμε να ξεπεράσουμε και να ξεπεράσουμε με την καλή πρόθεση όλων αλλά και με την ε, πεποίθηση και εκ μέρους του Κοινοβουλίου βεβαίως ότι αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη μας και ένα από αυτά είναι το ότι εάν η συνθήκη Λισαβόνας προσδίδει αυτή τη σημασία στο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτό οφείλεται κυρίως στην συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέδεσε τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αυτές τις δραστηριότητες. Η παρουσία και ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν προήλθε ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε προήλθε από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Απλά και μόνο γεννάται από την πεποίθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε πράγματι η, η οικοδόμηση που κάνουμε η ένωση που κάνουμε είναι μια ένωση με την οποία ταυτίζονται και στην οποία εκπροσωπώνται όλοι οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε σαφές το γεγονό ότι η δημοκρατική πρόοδος, η πρόοδος του εκδημοκρατισμού που απετέλεσε η οικοδόμηση της Ευρώπης τα τελευταία 50 χρόνια προσμετράται με την αύξηση των αρμοδιοτήτων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέκτησε από συνθήκη σε συνθήκη. Και αυτό αποτελεί νομίζω τον πύχη υπολογισμού ή μετρήσεως του επίπεδου εκδημοκρατισμού που έχουμε και που με τις συνθήκες της Λισαβόνας βρίσκει ένα καινούριο μεγάλο άλμα. Θα πρέπει βεβαίως να χαιρετήσουμε και την ε, συμφορά και συμβολή της Κομισιόν σε αυτή τη διαδικασία και χαιρετίζω εδώ μέσω του Προέδρου την συνεισφορά αυτή. Κάτι το οποίο βεβαίως περιπλέκει τα πράγματα κάποια φορά, αλλά εδώ ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πρόκληση, ώστε αυτά τα περίπλοκα πράγματα, αυτές τις περίπλοκες διαδικασίες, να μεταφραστούν σε πρόοδο και μεγαλύτερη συμμετοχή στην διαδικασία αυτή όλων των πολιτών μας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκροτήσαμε μία αρμόδια ομάδα, η ομάδα καθοδήγησης της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε αυτή την ομάδα, ομάδα καθοδήγησης, προεδρεύω εγώ και αποτελείται από τους προέδρους των Επιτροπών του Κοινοβουλίου και εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου και οθετήσαμε ένα έγγραφο το οποίο εξάλλου εγκρίθηκε και από τα διευθύνοντα όργανα του Κοινοβουλίου έγγραφο το οποίο δεν είναι τυχαίο νομίζω αλλά είναι ένα έγγραφο έστω και αν είναι εσωτερικό έγγραφο είναι επίσημο και θεωρώ ότι ο καθένας από εσά θα έπρεπε να λάβει γνώση αυτού του εγγράφου επειδή αυτό το έγγραφο είναι γνωστό στις ε, διοικήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είμαι βέβαιο όμω ότι κανείς από εσά δεν γνωρίζει το έγγραφο αυτό και θα ήταν πολύ σημαντικό ο καθένα από εσά να έχει πρόσβαση στο έγγραφο αυτό και να λάβει γνώση των συλλογισμών που έχουμε στο Κοινοβούλιο, πού φτάσαμε, πού έχουμε φτάσει και πώς θα μπορούσε να υπάρξει η απαραίτητη εκλογήκευση αυτών των σχέσεών μας ώστε να φτάσουμε στην μέγιστη αποτελεσματικότητα και στην μέγιστη ροή και ρευστότητα όσον αφορά τις αρμοδιότητες των μεν και των δε. Νομίζω ότι στην σημερινή και τη χθεσινή συνεδρίαση είχαμε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα με κριτικές που ασκήσαμε κάποιοι για την έλλειψη ας πούμε παρουσίας, επαρκούς παρουσίας μελών της Ευρωβουλής. Αυτό θα πρέπει να το ρυθμίσουμε γιατί αυτές οι συναντήσεις που είναι τόσο σημαντικές και είναι και λίγες δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών ώστε να μην υπάρχουν εδώ διχασμοί να μην χρειάζεται δηλαδή εδώ να παραστεί κάποιος αλλά και ταυτόχρονα κάπου Πάντως είχαμε συνεισφορές και συμβολές οι οποίες αποτελούν πηγή έμπνευση όχι μόνο από το Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά και χθε ε, είχαμε την συμβολή του κυρίου Ζουαγέ το οποίο το κείμενο έχει διανεμηθεί και νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που μας είπε ο κύριος Ζουαγέ που μας είπε ότι δηλαδή χάρη εν μέρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξεπεράσει το χειρότερο σημείο της κρίσης και όπως είπε και ο πρόεδρος της Κομισιόν που το είπε έτσι με τριοφροσύνη είναι αλήθεια ότι δεν αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες την ίδια κατάσταση όσον αφορά την έξοδο από την κρίση. Σε κάποιες χώρες ήδη βλέπουμε ότι έχουν βγει από την κρίση και αρχίζουν να οικοδομούν το μέλλον τους. Σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι είναι βαθιά μέσα στην κρίση και έχουν μεγαλύτερες ανησυχίες για το πώς θα βγουν από την κρίση παρά για το τι θα κάνουν στο μέλλον. Έχουν δηλαδή περισσότερο άγχος για την έξω από την κρίση και ασχολούνται λιγότερο με την οικοδόμηση του μέλλοντός τους. Πάντως το μέλλον αυτό μας αφορά όλους και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον από τις τωρινές, από τις παρούσες προκλήσεις. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Νομίζω ότι κάποιες ιδέες που ανέκυψαν όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμενο, η Οικονομική Διακυβέρνηση, η Φορολογική Εναρμόνιση, το θέμα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, τα κοινωνικά τα θέματα, όλα αυτά τα θέματα ακόμα δεν έχουν προοδεύσει επαρκώς, αλλά νομίζω ότι με την κοινή μας προσπάθεια θα πετύχουμε κάποια πρόοδο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε και για την συμμετοχή σας. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας λοιπόν και βεβαίως να ευχαριστήσω την, ε, τον πρόεδρο της Κομισιόν που παρά το βιβαρημένο του πρόγραμμα αποφάσισε να έρθει εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, να τον τιμήσω. Ευχαριστώ πολύ Μανουέλ που ήσουν εδώ μαζί μας. Φίλοι και φίλες, σας ε, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και θα ήθελα να ζητήσω τους υπαλλήλου να στείλουν σε καθένα από εσά το έγγραφο αυτό της Κατευθυντήριας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει και τόσο το έγγραφο αυτό να φτάσει στην διοίκηση των Εθνικών Κοινοβουλίων, που εκεί θα να, εκεί θα έπρεπε να πάει και να μείνει σε ένα, σε σιρτάρι. Αλλά θα πρέπει συγκεκριμένα να πάει στους προέδρους των, των κοινοβουλίων των εθνικών γιατί πολλές φορές αυτοί έχουν να κάνουν βέβαια και άλλα πράγματα, είναι απασχολημένοι αλλά θα πρέπει να το δουν αυτό το έγγραφο θα πρέπει λοιπόν όλοι σας να λάβετε γνώση αυτής της εμπειρίας θα δείτε το έγγραφο αυτό αυτό οκτασέλιδο είναι χρήσιμο και θα ήθελα μετά να μου σχολιάσετε ό,τι σας απασχολεί σχόλια και παρατήσεις τις οποίες θα δεχτούμε με μεγάλη χαρά. Και με χαρά λοιπόν σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στις ε, πατρίδες σας. Ευχαριστώ πολύ.